Καλημέρα σας και χαίρομαι που είσαστε εδώ όλοι στις 9 το πρωί στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλημέρα σας και θα ήθελα να σας πω ότι θα μιλήσω αργά σήμερα. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί έχουμε όλες τις γλώσσες σήμερα εκτός από τα κρατικά και τα ελληνικά. Έχουμε και μια ομάδα επισκεπτών της κυρίας Σάντερ, 12 επιχειρηματίες της Federation Νασιονάλ, de Ελπίζω σωστά να τα προφέρω όλα αυτά. Και προγραμματίζουμε λοιπόν σήμερα την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Επασχόλησης. Ας μην καθυστερήσουμε άλλο. Θέλουμε να τελειώσουμε λοιπόν ε, στις 12.30 ε, και μετά... Α, έχουμε μόνο μία ώρα λοιπόν τώρα στη διαθέσή μας. Ε, τώρα τα πρακτικά λοιπόν τις 16ης και 17ης ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις, αν όχι. Να περάσουμε στο σημείο 4, στο Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2017. Όλα τα τμήματα. Και θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον Γιάννη Γκάιερ, ο οποίος είναι αρμόδιος εισηγητής για φυγανικό αυτό προπολογισμό και ο συνάδελφος Γκάιερ όμως πρέπει να σας πω ότι κάπου έχει κολλήσει στην κίνηση. Δεν προχωράει. Και γι' αυτό λοιπόν δεν έχω και πολλά να σας πω. Γιατί για το σημείο αυτό ε, δεν μπορούμε να πάρουμε και στο επόμενο σημείο, γιατί θα μπλεχτούν τα υπόλοιπα και τα επόμενα θέματα. Και εγώ ο ίδιος ε, δεν μπορώ να σας παρουσιάσω την έκθεση του κυρίου Γκάιερ, γιατί θα με παρεξηγούσε κιόλα. Την κατανόησή σας λοιπόν ζητώ να περιμένουμε μέχρι ότου καταφτάσει ο συνάδελφος Γκάιερ και θα κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διάλειμμα. Αλλά σας παρακαλώ, οι λίγοι και έκλεκτοι που έχουν έρθει να μείνουν στην αίθουσα, γιατί σε λίγο μπορεί να είμαστε ακόμα λιγότεροι. peut pas faire le point 5 en attendant? Non? Μήπως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με το 5 περιμένοντας παρακαλώ. Ja, wir haben, wir haben keinen der heute Vormittag vorgesehenen Berichterstatter zur Verfügung, außer mir. Wir können den Tagesordnungspunkt 5. Κα, κα, κανείς από τους εισηγητές που έχουμε προβλέψει ε, μέχρι τώρα δεν έχει έρθει, οπότε ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με το 5. Εδώ είναι η κυρία Σαρτιέ βέβαια και κάποιοι άλλοι σκιώδεις, αλλά πολλοί άλλοι σκιώδεις ε, λείπουν. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να κάνουμε μία συζήτηση. Και από ό,τι φαίνεται ο εισηγητής για το πρώτο θέμα, για το σημείο 4 της σημερινής διατάξης, ε, κατέφτασε, καταφτάνει. Also kann sich's nur noch um So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem nun... Αγαπητοί συνάδελφοι, τα κατάφερε να απελευθερωθεί από την πρωινή κίνηση ο κύριος Γκάιερ με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί οτιδήποτε λιγότερο από μισή ώρα είναι μικρή καθυστέρηση. Μπορούμε λοιπόν πάρα αυτά να ξεκινήσουμε στο σημείο 4, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2017, όλα τα τμήματα. Και να καλωσορίσω λοιπόν τον εισηγητή Γιένς Γκάιρ, εισηγητή χωρίς ε, ε, να μακρηγορήσω. Θα του δώσω το λόγο για να μην χάσουμε κι άλλο χρόνο. Λοιπόν, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους για την καθυστέρηση την οποία υπέστησα, γιατί κανονικά φεύγω στις 8.30 για το Κοινοβούλιο, αλλά σήμερα διαπίστωσα ότι τα πράγματα έχουν χειροτρέψει στην κίνηση σε αυτή την πόλη και ληστώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Μπαίνω λίγο στον πειρασμό να σα πω ότι θα μιλήσω πιο γρήγορα, αλλά να με δυσκολέψω για τη τερμηνείς. Ε, να είμαι λοιπόν όσο πιο συγκεκριμένο γίνεται. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον προπολογισμό για το 2017, βρισκόμαστε στο σημείο όπου αναμένουμε δημοσίευση του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 25 Μαΐου. Και μετά θα ξεκινήσουμε τις εργασίες μας επί του σχεδίου αυτού. Επί της διαδικασίας, εν συντομία, να σας πω το εξή ότι καταρχάς το σχέδιο προϋπολογισμού θα διαβιβαστεί προς το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα επεξεργαστεί βάσει των κρατηντρίων γραμμών του το σχέδιο προϋπολογισμού να κάνω μια μικρή παρένθεση και μια προσωπική εκτίμηση να σας δώσω και το συνέχεια το, το Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί το τροποποιημένο σχέδιο προπολογισμού από το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη ολομέλεια του Στρασβούργου αποφάσισε επί των δικών του κατευθυντηρίων γραμμών. Και χαίρομαι που το μεγαλύτερο τμήμα του Κοινοβουλίου ακολούθησε η μεγάλη πλειοψηφία του Κοινοβουλίου την πρότασή μου, όπως τροποποιήθηκε και από τις προτάσεις των συναδέλφων. Σε ό,τι αφορά τώρα το Συμβούλιο, θεωρώ ότι το Συμβούλιο είναι business as usual, ακολουθεί λίγο το, αυτά που έκανε τα τελευταία χρόνια, ενώ το Κοινοβούλιο ενασχολείται κάπως πιο σοβαρά με τον προπολογισμό. Για τον τρέχοντα λοιπόν προπολογισμό, το 2016, αγαπητοί συνάδελφοι, στην κατηγορία 3, εσωτερική πολιτική, και στην κατηγορία 4, εξωτερική πολιτική, έχουμε τα περιθώρια τα οποία έχει θέσει το Μεσοπρόθεσμο Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα όρια δηλαδή σε ό,τι αφορά τις δαπάνες στις κατηγορίες αυτές, έχουν ε, εξαντληθεί πλήρως μετά την προσφυγική κρίση. Άρα, ως εκ τούτου, στην κατηγορία 4, στην εξωτερική πολιτική, έχουμε κινητοποιήσει όλους τους πόρους για να καταπολεμήσουμε τους λόγους προσφυγίας, για την υποστήριξη της Συρίας στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, για την παροχή τροφίμων, για τους πρόσφυγες, για την εκπαίδευση των παιδιών και όλα αυτά και στην κατηγορία 3 το ίδιο έχει γίνει σε ό,τι αφορά τον Ταμείο για το άσυλο και την ε, μετανάστευση και με εργαλεία τα οποία ως σκοπό έχουν να ενισχύσουν τα κράτη-μέλη στην ε, διαφύλαξη των συνόρων. Με το σύστημα των ανοιχτών συνόρων προκειμένου να διαχειριστούν το σύνορά του όσο πιο καλά γίνεται με τα περιορισμένα μέσα που έχουμε. Το Συμβούλιο λοιπόν όλα αυτά δεν τα παίρνει υπόψη. Και όταν διάβασα τι κατευθυντήριε γραμμέ, εγώ νόμιζα ότι μπερδεύτηκα. Ε, και ότι πήρε το έγγραφο τη περσινή χρονιά. Γιατί στα πρώτα, στι πρώτε τέσσερι σελίδε ε, είχαν αλλάξει μια μισή φράση μόνο. Και κατά τα άλλα ήταν το ίδιο κείμενο όπω πέρσι. Μόνο τι δύο τελευταίε σελίδε είχαν αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Σας παρακαλούμε μην εξαντλείται τις δαπάνες μέχρι το ανώτατο όριο, γιατί θέλουμε περιθώριο ελιγμού σε περίπτωση αναπάντεχων περιστατικών. Αυτό είναι το ζουμί του Συμβουλίου. Εγώ, αγαπητοί συναδελφοί, δεν ε, βλέπω οποιαδήποτε, οποιοδήποτε λόγο για τον οποίο θα μπορούσε να έχει αλλάξει κάποια από τις ε, κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε διαφορετική στάση, να έχουμε διαφορετική στάση το 2017. Όλοι προφανώς ελπίζουμε να βελτιωθεί η κατάσταση στη Συρία, να ερεμίζουν τα πράγματα, ενδεχομένως να πάμε και σε κατάπαυση πυρός, να οδηγηθούμε ενδεχομένως πάλι σε μια ερνευτική διαδικασία η οποία θα οδηγούσε τον κόσμο να επιστρέψει στην πατρίδα του για να την ανοικοδομήσει, αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Και άρα τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε φέτο για την αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση. θεωρώ ότι θα τα χρειαζόμαστε και στη συνέχεια και στο μέλλον. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα τμήμα τη αντιπαράθεση που θα έχουμε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία έγκριση του προπολογισμού. Η οικονομική κατάσταση έχει βελτιωθεί σε κάποιες ε, χώρες αλλά στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, έχουμε μεγάλα, μεγάλη απόσταση να καλύψουμε. 8 δις πρέπει να βγάλουμε από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για να υπάρχει εγγύηση και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις από πλευράς του ΕΦΣΥ. 3,8 δις είχαμε ως τώρα. Άρα έχουμε μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλη δυσκολία τα πού θα βρούμε τα χρήματα για να συμπληρώσουμε το Ταμείο ΕΦΣΥ. Και άρα ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε απόλυτα τα εργαλεία του προϋπολογισμού, τα μέσα του προϋπολογισμού και να συνεχιστεί η πολιτική δέσμευση και προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή για να υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υπεραξία δε στις δαπάνες, προτείναμε στις κατευθυντηρίες γραμμές τα μέσα του προϋπολογισμού που δαπανούμε για την κατηγορία 1α, 1β κυρίως, να στραφούν και να συνδεθούν με τις οικονομικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πιο σαφή τρόπο υπάρχει ε, το έγγραφο των οικονομικών προοπτικών σε ό,τι αφορά το 2015. Υπάρχει η ετήσια αναπτυξιακή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο υποδεικνύει το ποιε δομέ και υποδομέ θα πρέπει να αλλάξουν στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι κατευθυντήριε γραμμέ για το πώ ε, θα υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει ότι θα υιοθετήσουμε ε, άκρητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κοινοβούλιο, αλλά ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία για να δούμε κατά πόσον υπάρχει στοχευμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο αυτή η προσέγγιση για να υπάρχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή υπεραξία. Αυτά, συνάδελφοι, και μέσα σε όλα αυτά προφανώς συνεχίζονται και τα σημεία προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, του παρελθόντος. Ε, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Είχαμε αφήσει ένα κενό εδώ, γιατί είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχά να αξιολογηθεί η κατάσταση τη ευρωπαϊκής αυτή Πρωτοβουλία για την νεολαία και μετά να δούμε κατά πόσο τα πράγματα κινούνται προ την κατεύθυνση που επιθυμούσαμε. Δεν ε, συμφώνησε τα τελευταία χρόνια απαραίτητα με την πρόταση αυτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε ποια θα είναι η εκτίμηση και η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε τι θα συνεπάγεται αυτό και σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες. Θέλουμε επίσης να συνεχιστεί η καταπολέμηση της ένδυας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τμήμα της στρατηγικής της Ευρώπης το 2020 και το πρότασή μου ήταν να φροντίσουμε να θέσουμε στο επίκεντρο την καταπολέμηση της ε, φτώχειας ε, για τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά τις απληρωμές, πλέον ε, δεν έχουμε μεγάλο κύμα απλήρωτων λογαριασμών, δεν έχουμε φυσικά εκπληρώσει όλες μας τις υποχρεώσεις. Άλλα τα πράγματα πάνε καλύτερα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτική. Έχει να κάνει κυρίως με τι χρηματοοικονομικέ ροέ. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, να σας το εξηγήσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι καθοριστικό αυτό για τη σημερινή συζήτηση. Να επισημάνω μόνο ότι δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα πλέον σε ό,τι αφορά τους απλήρωτους λογαριασμούς, αλλά όλοι οι ειδικοί σε θέματα προϋπολογισμού φοβούμαστε ότι αυτό θα επανέλθει, αλλά εν περιπτώσει δεν μας επιβαρύνει για τον προπολογισμό του 2017, Αυτές είναι λοιπόν οι γενικότερες συνθήκες, οι γενικότεροι όροι ε, μέσα στους οποίους θα πρέπει να εργαστούμε και με χαρά μου θα ακούσω τα σχόλια των συναντέλφων από την Επιτροπή Επασχόλησης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα να ξεκινήσουμε κατευθείαν τη συζήτηση με τους σκιώδεις. Από το ΕΛΚ το λόγο έχει... Μάλλον δεν ε, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος. Η Ελίζα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και στον εισηγητή του προπολογισμού που μας έδωσε την εικόνα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα ειλικρινής και ρεαλιστική εικόνα αυτή. Λοιπόν, μέσα στην κατάσταση που μας περιγράψατε βλέπω ότι τώρα είναι η ώρα, ή ποτέ, όπου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις θέσεις του σε σχέση με την ε, βούληση ή την έλλειψη βούλησης από πλευράς ε, του Συμβουλίου. Σας στηρίζουμε λοιπόν πλήρως αυτό. Δεν ε, μπορούμε να βασιζόμαστε σε κάποιες αρχές business as usual, όπως είπατε και εσείς πριν, γιατί οι καταστάσεις έχουν αλλάξει και οποιαδήποτε διατάραξη της ισορροπίας θα πρέπει να προβλέπεται στον προπολογισμό. Αυτό είναι που με απασχολεί, αυτό είναι που απασχολεί γενικότερα την Επιτροπή μας, αλλά φαντάζομαι και όλους τους συναδέρφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από όποια πολιτική ομάδα και αν προέρχονται. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε όπως κάναμε παλιότερα με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς, γιατί η τεράστια μετακίνηση προσφύγων αλλά και η μετανάστευση έχει τροποποίησει τις ανάγκες και τις απαντήσεις που καλούμεθα να δώσουμε στις νέες αυτές ανάγκες. Το να συνεχίζουμε να λέμε αφήστε τα περιθώρια, μην τα χρησιμοποιείτε, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να ακούμε κάτι τέτοιο πια. Και όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή μας Απασχόλησης, υπάρχει εδώ ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρο, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πάντα. Και αυτό είναι οι προθεσμίες για το 2017, αλλά επιπλέον έχουμε και την αναθεώρηση των πολιετών ε, πολιτικών μας στα μέσα της περίοδου. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι μέσα έχουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Τι μας απασχολεί. Το κοινωνικό Ευρωπαϊκό Ταμείο, το οποίο αποτελεί τον μοχλό για την βελτίωση της απασχόλησης. Δεν είναι έτσι ένα τυχαίο εργαλείο. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι αυτή η οποία βοηθάει να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Άρα είναι απαραίτητο να το στηρίξουμε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επίσης, η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η εγγύηση για την νεολαία είναι η βάση, είναι η θεμελιώδης πολιτική, ουσιαστική. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι αυτό που θέλουν να περνάνε στον κόσμο κάποιοι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά η πραγματική πολιτική του Ταμείου, αυτή η οποία θα επιτρέψει, όπω είπατε, να καταπολεμήσουμε την φτώχεια των παιδιών, είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των γονιών του. Άρα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Και σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η εγγύηση για την νεολαία. Αυτό στηρίζουμε. Και αν θέλουμε να υπάρξει και επαγγελματική αποκατάσταση των ε, προσφύγων μετά από πιστοποίηση των διπλωμάτων, τους ε, ισοτιμιών κτλ. Δεν θα βρούμε τα χρήματα στο περιθώριο γιατί θα είναι μια πραγματική πολιτική. Άρα, επ' αυτού, εγώ κινητοποιούμε και να ξέρετε ότι το ΕΛΚΑ στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα δώσει μεγάλη σημασία σε αυτήν την πολιτική επαγγελματικής ένταξης για να είναι αποτελεσματική. Γιατί καταλαβαίνετε, το θέμα δεν είναι να επιδοτούμε, να βοηθάμε. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι πατερίτσες. Αυτό το κάνουμε όταν έχουμε αποτύχει αλλού. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια πραγματική επαγγελματική ένταξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πυρίνσκι τώρα από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γκάιερ και η κυρία Σαρκή. Τα πράγματα δεν είναι απλά κανονικά και συνηθισμένα αυτή τη φορά. Να μου επιτρέψετε λοιπόν κύριε Πρόεδρε εδώ να εκφράσω την βαθύτατη μου ανησυχία λέμε ότι τα πράγματα είναι έκτακτα, χρήζουν έκτακτης αντιμετώπισης, αλλά παρόλα αυτά δεν κάνουμε τίποτα. Και το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα όργανα έχουν ας πούμε συζητήσει το θέμα της ασφάλειας των συνόρων. Έχουν συζητήσει διαφορετικές ρυθμίσεις για μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιεί και το μαστίγιο και το καρότο σε θέματα που άπτονται στην άμυνά της και την ασφάλειά της. Η κοινωνική πόρη και η απασχόληση έχει άμεση σχέση με το επίπεδο ασφάλειας το οποίο ζούμε στην Ένωση και στην γειτονική περιοχή. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πάνω σε αυτό. Να πω όμως ότι η κοινοβουλευτική μας επιτροπή θα πρέπει να παίζει ηγετικό ρόλο στη συζήτηση στο Κοινοβούλιο γύρω από το θέμα αυτό και να διαμορφώσει τη θέση του Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο. Το οποίο ακολουθεί διαφορετικές προοπτικές και δεν καλύπτει τις ανησυχίες μας. Τώρα για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό το παιχνίδι του κόβω και ράβω, δηλαδή κόβω λίγο από εδώ και προσπαθώ να τα αναπληρώσω από αλλού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, δεν είναι σοβαρή λύση. Αυτά τα οποία προτείνονται και γίνονται δεκτά πρέπει να επιβεβαιούνται και να μην υπάρχει μια μόνιμη αμφιβολία για το τι θα συμβεί στις διαπραγματεύσεις. και για το θέμα της κάλυψης των αναγκών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Υπάρχει η αίσθηση ότι το 2016 θα υπάρξει υπερβολική πίεση απαιτήσεων από το κοινωνικό ταμείο. Και θα πρέπει να υπάρξουν πάρα πολλές πληρωμές και στο τέλος του 16 και το 17 και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε Και αυτό έχει σημασία και με το σημείο 5 για τον τριγωνικό διάλογο που θα συζητήσουμε. Τώρα για το Ταμείο για την ακραία φτώχεια είναι σαφές ότι θα πρέπει να καλυφθεί σε επίπεδο πιστώσεων. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα της εγγύησης, του μέσου εγγύησης για τους νέους, για την καταπολέμηση της φτώχειας των παιδιών. Και όπως είπε ο Χανς Γκάια, υπάρχει και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου, που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για το τρίτο τμήμα και στην παράγραφο 12 και 13 υπάρχουν σαφέστατες προβλέψεις και ρήτρε για το τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις κοινοβουλευτικές μας προτεραιότητες. Ο Γένς αναφέρθηκε και στον κίνδυνο που υπάρχει για ε, ε, μια άλλη σώρευση καθυστερημένων και απλήρωτων υποχρεώσεων ε, που θα πρέπει κανονικά να μην υπήρχε το 2017. Και σχετικά με τα ειδικά μέσα, τώρα όπως ε, η αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και η κάλυψη των οικονομικών αναγκών του Ταμείου αυτού, θα πρέπει να ξεπερνούν το επίπεδο του MFF, όπως γίνεται και με τις υποχρεώσεις είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε στην ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και για το 2017. Όπως αυξάνουμε τις πιστώσεις υποχρεώσεων, έτσι θα πρέπει να αυξήσουμε και τις πιστώσεις πληρωμών. Τώρα, για τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε καλύτερα τα επιχείρηματά μας. η σοσιαλιστική ομάδα επιφυλάσσεται και θα καταθέσει νέες προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Ε, η κ. από το ECR. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εισηγητή. Γιατί ο κύριος Γκάιερ το επεσήμανε και ο ίδιος ότι περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και αυτό στην παρέμβαση φάση μας αναγκάζει να κάνουμε μόνο γενικά σχόλια. Κύριε πρέπει να μιλήσω αν δεν Κύριε Μπρόκ, επιτρέψτε μου να πάρω το λόγο. Σχόλια εκτός μικροφώνου του κυρίου Μπρόκ. Η πρόταση λοιπόν του εισηγητή περιλαμβάνει ε, διάφορες αξιώσεις για προγράμματα, αλλά δεν ε, βλέπω προτάσεις για το πώς μπορούμε να ανταπανίσουμε αποτελεσματικά τα, τους φόρου. Ε, φόρους, τους πόρους. Μία από τις βασικές αρχές ήταν ε, η αρχή της υπεραξίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό ένα ευρωπαϊκό μέτρο από το αντίστοιχο ε, περιφερειακό, τοπικό μέτρο. Και θα θέλαμε λοιπόν κατεπηγόντως να κρατήσει το Κοινοβούλιο αυτό ως κατευθυντήρια γραμμή, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε υποστήριξη και από τους πολίτες. Συγκεκριμένα, πιστεύουμε για παράδειγμα ότι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως, ε, από προγράμματα όπως το COSME είναι πάρα πολύ καλά Χρειάζεται μια καλή αξιολόγηση και θα έπρεπε αυτή η αξιολόγηση να αποτελεί προϋπόθεση για την δαπάνη πόνων. Στα κοινωνικά και στα θέματα απασχόλησης, για παράδειγμα η πρωτοβουλία για την, ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αναφέρθηκε και για τον εισηγητή. Εδώ θα ήθελα να προτείνω το εξή. Κατεπηγόντως να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού, θα πανηθούν περαιτέρω πόροι. Επίσης, ο εισηγητή φυσικά επεσήμανε και το θέμα της καταπολέμησης της στόχιας και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά της παιδική ένδυας. Πώς να το... να μην το υποστρίξουμε αυτό ως στόχο, αλλά δεν είναι σαφές τι γραφειοκρατία συνεπάγεται αυτό και πώς πρέπει να το υποστηρίξουμε. Θέλω μεγαλύτερη σαφήνεια. Και τέλος, ε, ε, Ακούσαμε και την προσφυγική κρίση. Για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης θα θέλαμε να χρησιμοποιηθούν και πόροι από το ε, Ταμείο Συνδρομής για τους ε, λιγότερο, για τους πιο μειονεκτούντες, ε, τα, πιο, τα με τα μειονεκτήματα στον πληθυσμό, γιατί ως τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χόπκιν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε σήμερα το πρωί και για τις προοπτικές που μας παρουσίασε. Ε, δεν θα διαφωνούσα με τα όσα άκουσα μέχρι τώρα. Εντάξει, συνολικά πράγματι όλα έχουν αλλάξει. Όλοι το λένε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όμως αυτό που προσπαθώ εδώ να δω είναι τι συγκεκριμένα βήματα μπορούμε να αναλάβουμε για να μην συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα σαν να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Συμφωνώ με τον κύριο Πυρίνσκι όταν είπε ότι υπάρχει στον προπολογισμό, υπάρχει, δεν πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Αυτό είναι σπατάλη χρόνου και ενέργειας. Αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό που χρειάζεται είναι κάποια ριζοσπαστική αλλαγή, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζοσπαστικά βρίσκεται στο ριό του προπολογισμό και η προσφυγική κρίση έχει πολλέ επιπτώσει. Μία από αυτέ είναι στον προπολογισμό. Και ο προπολογισμό δεν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Η κυρία Σαρτιέ επίση έχει δίκιο ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που ήδη διαθέτουμε, όπω είναι το Φεντέρο, όπω είναι το Κοινωνικό Ταμείο. Είναι πράγματα που θα βοηθήσουν, αλλά κατά τη γνώμη μου η χρηματοδότηση δεν είναι επαρκή. Άρα χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Και έχουμε αναλάβει πολλές δεσμεύσεις, οπότε η... ο βαθμός ευελιξίας που διαθέτει σήμερα ο προπολογισμό δεν φτάνει. Εδώ λιγάκι τα λέω στον εαυτό μου. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να βρούμε τρόπο ώστε σε 12 μήνες που θα ξανάρθουμε εδώ να πούμε καταφέραμε να κάνουμε το α, το β και το γ. Ούτε εγώ το έχω ξεκάθαρο στο κεφάλι μου. Γι' αυτό και θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέρφων επ' αυτού. Ο εισηγητής είπε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε ότι πρέπει τα ταμεία να τα χρησιμοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο, στοχοθετημένα. Οπότε πράγματι, ας δούμε πού δαπανάμε τα χρήματα και να είμαστε σίγουροι ότι τα δαπανάμε με έξυπνο τρόπο, φροντίζοντας να υπάρχει πάντα προστιθέμενη αξία. Μετά θα συζητήσουμε για την εντολή για τον τριημερή διάλογο και τα υπόλοιπα θα τα πω τότε. Για αυτό το θέμα αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους. Δεν έχω εισηγητή καταγεγραμμένο. Ούτε ζητάει και το λόγο. Η δεν έχει ορίσει και αυτή η ε, εισηγητή και η κυρία Μητσότα θα ήταν η επόμενη, αλλά και αυτή δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνηθισμένα πράγματα αυτά που είπατε. Εντυπωσιάστηκα όμως από αυτά τα οποία είπε ο Γενικός Συγητής. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω Βέβαια προκαλούν φόβο αυτά που ακούσαμε. Η λογική του business as usual φοβάμαι ότι δεν θα αποδώσει. Κάνουμε τα πάντα και δεν κάνουμε τίποτα. Είπατε και το ξέραμε βέβαια ότι στην κατηγορία, στην κατηγορία 3 και στην κατηγορία 4 οι πιστώσεις στο τέλος Απριλίου έχουν ήδη εξαντληθεί λόγω της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. τι θα γίνει με την υπόλοιπη περίοδο λοιπόν. Θα σεβαστούμε τις υποχρεώσεις ή θα πρέπει να πάρουμε τα χρήματα από άλλες γραμμές για να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Έχει σημασία αυτό που λέτε ότι οι πολιτικές μας υπέρ της απασχόλησης των νόεων ε, δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικές είναι. Καιρός ήταν να το αναρωτηθούμε αυτό. Πέρα από το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να καθορίσει τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στα πλαίσια και των στόχων 2020. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η κυρία Μωρέν Σαρτιέ. Για να κλείσω και να μην σας καθυστερώ, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Γκάιερ μας περιγράφει τη δημοσιονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πίθο των Δαναίδων. Δεν ξέρουμε τι βάζουμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι βγάζουμε από τον πίθο των Δαναίδων. στην ουσία περιμένει να υπάρξουν πάρα πολλές ακάλυπτες υποχρεώσεις. Στην ουσία προετοιμάζουμε τον προϋπολογισμό του 17 έχοντας στη διάθεσή μας τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή μας το 14. Ή μήπω αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε και συζητάμε τη μελλοντική μας πτώχευση. Κάνετε διάφορες παρατηρήσεις για τη φτώχεια, τη δυστυχία, την ένταξη, την κοινωνική μέσω της εργασίας. Φοβάμαι ότι όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρό τρόπο και όλα αυτά έχουν έναν λόγο και ο λόγος αυτός είναι το κοινωνικό dumping. Να σας θυμίσω την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, για την απόλυτα ελεύθερη μορφή του ανταγωνισμού και εδώ ίσως ο Πρόεδρος να συμφωνήσει λίγο μαζί μου. Οι εμπορικές συμφωνίες μήπως που ετοιμάζουμε, το TTIP, όλα αυτά φοβάμαι ότι αγνοούνται από τον εισηγητή του προϋπολογισμού και αυτά είναι τα προβλήματα. Να μην μιλήσω τώρα για τον έλεγχο των συνόρων και τα λοιπά, ξέρετε ποια είναι η άποψή μας. Επαναλαμβάνω εμείς δεν έχουμε τα μέσα για να υποδεχθούμε τη δυστυχία του κόσμου όλου και υπάρχουν άλλες χώρες κοντά στη Συρία να τους υποδεχτούν. Γιατί πρέπει να το κάνει η Ευρώπη μόνο ξανά και ξανά. Λοιπόν, αν πράγματι θέλουμε κάτι να κάνουμε, είναι να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες να βγάλουμε θέσεις δουλειάς. Ο κόσμος όταν δουλεύει έχει αγοραστική ικανότητα, μπορεί να σπουδάζει τα παιδιά του, και το 80-80 με 90% των ανθρώπων που εργάζονται, εργάζονται στις μικρομεσαίες. Βοηθήστε τις μικρομεσαίες να προσλάβουν και να επαναπροσλάβουν. Μάλιστα και εγώ θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποια δικά μου σχόλια, να προσθέσω τα δικά μου σχόλια. Ο εισηγητής ε, μας είπε ότι τις επόμενες ημέρες κάποια στιγμή θα λάβουμε και την αξιολόγηση για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και ελπίζω ιδιαίτερα να μην μας παρουσιαστεί η παρουσίαση αυτή, η αξιολόγηση αυτή όπως αποτελεκτικό συνέδριο για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης της Νέους γιατί ήταν ε, καλό αυτό το σχέδιο, αλλά από ό,τι φαίνεται κόλλησε στα περαιτέρω, στη γραφειοκρατία. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την ε, προώθηση της απασχόλησης των νέων. Και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Γκάιερ για να κλείσει. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η κυρία Χόκκιν για το τι χρειάζονται, κατά πόσο χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές και τι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα να κάνουμε βήμα πίσω. Καλώς όρισα έντερμα την ε, συνθήκη της Λισαβόνα. Θεωρώ μόνο ότι ένα πρόβλημα υπήρχε με τη συνθήκη της Λισαβόνα από πλευράς του προϋπολογισμού και των υπεύθυνων προϋπολογισμού. Έχουμε στον προϋπολογισμό μία μόνο ανάγνωση και αυτό από κοινοβουλευτικό επίπεδο μας αποδυναμώνει σε σχέση με την κατάσταση προ-Λισαβόνας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μία κατάσταση όπου πρέπει να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Και όσο κι αν με πονάει, δεν θέλω να έχουμε και αυτά σε ό,τι αφορά τη θέση μας στην διαπραγματευσή αυτή. Δεν θέλω να υποκρινόμαστε ότι είμαστε πιο δυνατοί από ότι είμαστε στην ουσία. Μην δίνουμε λάθος εντυπώσεις. Το κλειδί για την επιτυχία των διαπραγματεύσεων ήταν η Προεδρία. Και αυτό δυστυχώς ήταν ε, καταστροφικό υπό την Ιταλική Προεδρία, πάρα πολύ καλό υπό την Λουξεμβουργιανή Προεδρία που προσπάθησε να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο και τελικά καταλήξαμε σε μια συμβουλευτική θέση η οποία υποστηριχθήκε και από τι δύο πλευρές. Αν τώρα στην καθοριστική φάση των διαπραγματεύσεων ε, ε, με την... Στη, μάλλον στην καθοριστική φάση των διαπραγματεύσεων θα είμαστε με την ε, Σλοβακική κυβέρνηση. Και θα συνδεθώ σήμερα το βράδυ μαζί τους μάλιστα με εκπροσώπους τους για να δούμε πώς θα γίνει τεχνικός πώς αυτή η διαπραγμάτευση. Η Ιταλική Προεδρία πέρσι άφησε να περάσουν δύο εβδομάδες, μετά κατέληξε σε συμφωνία στο Συμβούλιο και μετά ήρθε στο Κοινοβούλιο και μας είπε να, αυτό πρέπει να εγκρίνεται. Αυτό λοιπόν ήταν τόσο ευαίσθητο και ήταν τόσο ευαίσθητε οι ισορροπίε μεταξύ των κρατών μελών που δεν καταφέραμε να κάνουμε και τίποτε. Θα δω λοιπόν πώ θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Θα δω πώ θα τα πάμε και με την σλοβακική κυβέρνηση. Στη φάση αυτή δεν είμαστε τόσο δυνατοί όσο ήταν το κοινοβούλιο πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας, επαναλαμβάνω. Και βλέπω και συχνά ότι δεν το έχουν κατανοήσει πολλοί συνάδελφοι και πολύ υψηλή αξία το μαθητούχη της Επιτροπής δεν το έχουν κατανοήσει αυτό. Ύστερα, δεν ε, μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα και πόρους από κατηγορία σε κατηγορία. Δηλαδή, αν εγώ θεωρώ ότι κάποια κατηγορία έχει πολλούς πόρου. δεν μπορούμε να τις μεταφέρω κάπου αλλού, για παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το τρίτο σημείο τώρα, επί το περιεχομένου. Έχουμε μεγάλο περιθώριο στο τι μπορούμε να κάνουμε με τους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά αυτό ορίζεται ουσιαστικά στις ε, οδηγίες πλαίσιο σε ό,τι αφορά το, τους πόρους, για παράδειγμα, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό που μπορούμε να καθορίσουμε είναι το τι θα δαπανηθεί και σε ποια χρονιά και αυτό είναι που μας απασχολεί. Γι' αυτό τσακωνόμαστε, γι' αυτό σας είπα ότι το Συμβούλιο συνέχεια μας λέει ότι θα πρέπει να έχουμε όσο μεγαλύτερο περιθώριο γίνεται μεταξύ των ανώτατων πληρωμών και των ε, τρεχούσεων προβλεπόμενων ε, πληρωμών για να υπάρχει περιθώριο λιγμού. Και έτσι κάνει ε, εν μέρει αυθαίρετε σε περικοπές. Αυτή είναι η στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, αλλά θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Και αυτό για την κυρία Τριμπέζιους. Πάντα θέτει το θέμα τη σωστή αξιοποίηση των πόρων. Η επιχειρηματολογία είναι γνωστή από τους κόλπους του ECR και κάποιες φορές ε, στα γερμανικά, συνήθως στα αγγλικά. 80% αγαπητοί συνάδελφοι των δαπανών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δίδονται για έξοδο διαχείρισης. Δηλαδή τα κράτη-μέλη αποφασίζουν το πώς δαπανούνται τα οι πόροι του Περιφερειακού Ταμείου, για παράδειγμα. Το κατά πόσον ε, θα υπάρξει δηλαδή υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα χρήματα αυτά. Αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Και συνήθως τα κράτη-μέλη αποφασίζουν το πώς θα δαπανούν τα χρήματα στις περιφερειές τους και στις επικρατείες τους. Σωστό αυτό, αλλά αν 80% δαπανάτε για έξοδα διαχείρισης, αυτό ω ευθύνη βαρύνει του Δήμου και τι κοινότητε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και αν λοιπόν παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σωστή αξιοποίηση των πόρων, να στρέψετε την κριτική αυτή προ ε, τα μελη Οι Βρετανοί του ECR συχνά παραπονιούνται ότι δεν ε, δαπανώνται σωστά αυτή οι πόροι. Και θα αναφέρω το Ευρωπαϊκό Ρεκτικό Συνέδριο, άμα επιτρέπετε, που κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους για την δαπάνη των πόρων ε, στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, είναι ενδιαφέρον ότι το δεν τα πηγαίνει καλά το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Και κοιτώντα πώ θα πάνε, για παράδειγμα, οι πόροι για την αναπτύξη τη υπαίθρου ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπιστώνουμε, από το ελεγκτικό συνέδριο δηλαδή, ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων, μεγάλο τελεστή Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι αν δαπανούνταν καλύτερα αυτοί οι πόροι από τα κράτη-μέλη, αυτό θα ήταν πολύ καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν το κάνουν. Είναι λοιπόν περίπλοκα τα πράγματα αυτά. Σε ό,τι αφορά αυτό το ταμείο για τους πλέον ενδεείς. έχει προτεραιότητα, αλλά καταρχάς θα πρέπει να αποφασίσουν τα κρατημέλη κατά πόσον το θέλουν. Η Γερμανία δεν το υποστηρίζει και κατά πόσον θα εφαρμοστεί το ταμείο αυτό, κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί για τις πρόσφυγες. Αλλά καταρχάς εξαρτάται από τα κρατημέλη, όπως σας είπα. Και κατά δεύτερον, δεν είναι και πανάκια από Πλευρά ε, χρηματοδότησης. Είναι περιορισμένο το ταμείο αυτό. Άμα χρησιμοποιηθεί δε και για τους πρόσφυγες είναι γελία περιορισμένο το ποσό. Γιατί έχουμε 140 δις ό,τι αφορά το προπολογισμό των ευρωπαϊκό. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, καταλαβαίνετε δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Νομίζω όμως ότι όλοι θα αγωνιστούμε προκειμένου τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεση της η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανηθούν σωστά, αλλά πραγματική μόχλευση είναι στα περιφερειακά ταμεία, στα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης και εκεί θα πρέπει να μην είμαστε θύματα των αποφάσεων του Συμβουλίου, αλλά να προωθήσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει, όπως για παράδειγμα θέσεις απασχόλησης και όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να λυθούν σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχει το πλαίσιο, υπάρχει και ένα λειτουργικό πρόγραμμα και θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο τα πράγματα κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Ύστερα, ε, να πω ότι φυσικά και ξέρουμε πώς δαπανηθήκαν οι πόροι το 2014. Το ελεκτικό συνέδριο για αυτόν τον σκοπό την έκθεση του κάθε χρόνο. Και γι' αυτό κάνουμε και την έκθεση χορήγηση απαλλαγή σε ό,τι αφορά τα προγράμματα αυτά δαπανών. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο ε, επισταμένως είναι κατά πόσον υπήρξε ε, σωστό αποτέλεσμα, Σωστό αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τις μετέπειτα εξέλιξεις. Άρα, η Αντιπρόεδρος, η Γεωργίευα, ήθελε λοιπόν να θέσει στο επίκεντρο του προπολογισμού τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ένα προπολογισμό βάσει αποτελεσμάτων, αποδοτικότητα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει κάθε χρόνο. Θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο πολιετών προγραμμάτων, γιατί τα πιο πολλά προγράμματα είναι πολυετή. Καταρχά, λοιπόν, θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον η συμμόρφωση ήταν σωστή, κατά πόσον το πρόγραμμα απάντησε στα πραγματικά προβλήματα κτλ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς αγωνίζεται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, της δαπάνης των πόρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ συνάδελφε Γκάιρ, λέει ο Πρόεδρος, και νομίζω ότι η επόμενη τους επόμενους μήνες το θέμα του προϋπολογισμού θα μας απασχολήσει. Έχουμε διάφορα στάδια. Το πρώτο αναφέρεται και στο σημείο 5 του, της ημερησίας διάταξης σε ό,τι αφορά την ημερή διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό του κυρίου Γκάιερ. Σας ευχαριστώ. Άρα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης για τον προϋπολογισμό του 2017, εντολή για την έναρξη του ημερούς διαλόγου. Έχουμε ένα σχέδιο για την εντολή. Το σχεδίασε η γραμματεία. Δεν θα κάνω σχετικές αναφορές γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Είναι αρκετά σύντομο αυτό και αναφέρονται και διάφορα από την προηγούμενη συζήτηση. Θα πρέπει να επιμείνουμε για τον μελλοντικό προϋπολογισμό να προωθηθεί το πιο σημαντικό θέμα από πλευρά τη Επιτροπή Απασχόληση, το θέμα τη απασχόληση των νέων. Γι' αυτό λοιπόν και επιμένουμε στο θέμα αυτό και θα πρέπει να δούμε προκειμένου να υποστηριχθούν με αποτελεσματικό τρόπο τα προγράμματα αυτά. Και σε προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας αποφασίσαμε ότι σε κάθε περίπτωση θέλουμε να αποφύγουμε να δημιουργηθούν βουνά γράφων και πάλι. Άρα θέλουμε να υποστηρίξουμε πρακτικές λύσεις με τον προπολογισμό για τη δημιουργία καλών θέσεων απασχόλησης. Να επικεντρωθούμε στις ε, μειονεκτούσες αυτές ε, ομάδες στον τομέα της απασχόλησης, στους ε, πιο ηλικιωμένους, στους νέους, στους μετανάστες. και ότι κυρίω θέλουμε να υπάρχει μια καλή διαχείριση του προπολογισμού σε ό,τι αφορά τι εκθέσει του ελεκτικού συνεδρίου που μα παρουσιάστηκαν πριν από κάποιε εβδομάδε, σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για την νεολαία, για τα Youth Action Teams. Όλα αυτά κόλλησαν λόγω γραφειοκρατία κάπου. Αυτό δεν αποτελεί καλή ένδειξη σωστή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε τις δικές μας προτεραιότητες, χρειαζόμαστε δικές μας λύσεις και κυρίως λύσεις οι οποίες θα έχουν καλή χρηματοδότηση προκειμένου να τα πετύχουμε όλα αυτά. Ε, με ένα παράδειγμα να σας πω ότι εξηγώ. Εδώ και κάποιους ε, μήνες έχουν λάβει δύο πρωτοβουλίε. Η μία είναι μια διασυνοριακή εκπαιδευτική διαδικασία η οποία περνάει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ακούω από τους συζητητές ότι ναι, εντάξει, προχωρούν όλα αυτά, αλλά όταν στην πράξη θέλουμε να βρούμε ε, τι γίνεται, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ε, κάποια εφαρμογή. Δεν προχωράει, δεν κυλάει το, το ζήτημα, το πρόγραμμα. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει και το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να το βάλουμε στη συζήτηση είναι πώς θα δημιουργήσουμε τη σωστή υποστήριξη για την, την ένταξη των νέων μεταναστών. Όταν μιλάμε για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πάντα βγάζουμε κάποιες επικεφαλίδες, αλλά δεν θέλουμε συγκεκριμένα παραδείγματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, μπορούν να συνδεθούν με την απασχόληση των νέων, με την απασχόληση των νεαρών μεταναστών, που δεν έχουν ενδεχομένω ε, κάποια κατάρτιση, αλλά αν τους υποστηρίξουμε με ευρωπαϊκούς πόρους, Ενδεχομένως, να μπορεί να υπάρξει κατάρτιση των ε, νεαρών μεταναστών αλλά και των ε, επιχειρήσεων. Και αυτό θα έχει φυσικά αποτέλεσμα. Πέρσι να σας ότι δεν καλύφθηκαν α, ε, οι θέσεις απασχόλησης που προσφέρεται Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια σπατάλη πόρου σε ό,τι αφορά τα σχετικά προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν με τα προγράμματα αυτά να φροντίσουμε προκειμένου οι νεαροί άνεργοι, οι νεαροί μετανάστες, οι άνεργοι από χώρε όπου επικρατεί η οικονομική κρίση να προωθηθούν, να ενισχυθούν. Αυτό λοιπόν είναι ε, μια ιδέα η οποία ενδεχομένω να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκέ ε, γραμμέ. Σίγουρα λοιπόν θα μας απασχολήσει αυτό σε ό,τι αφορά τη συζήτησή μας ε, και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αυτά μέσα. Και αυτά θα πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί εδώ θα πληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Ευρωπαϊκός Προλογισμός. αν καθυστερήσουμε, αυτό δεν θα είναι καλή ένδειξη. Αυτά λοιπόν από δική μου πλευρά από το ΕΛΚ. Το λόγο έχει η κυρία Μωράν Σορτιέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την εντολή αυτή διαπραγματεύσεων εννοείται ότι έχετε όλοι μας την στήριξη. Και συνυπογράφουμε σε πολλά από αυτά που είπατε. Θέλω όμως να επανέλθω σε κάποια σημεία, τα οποία πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά. Τρία συγκεκριμένα. Πρώτον, η επαγγελματική ένταξη των νέων. Στις διαπραγματεύσεις, θα ήθελα, Πρόεδρε, στις διαπραγματεύσεις όπου θα πάτε και θα γηθείτε, θα ήθελα να είναι ξεκάθαρο ότι εμείς υποστηρίζουμε την εγγύηση για την νεολαία. Την ευρύτερη δηλαδή και την πιο θεμελιώδη πολιτική για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. Θυμίζω ότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων απλώς ε, ενισχύει την εγγύηση για την νεολαία, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία νέων. Αλλά μην κάνουμε εμείς ήδη, μην αυτοπυροβοληθούμε για τη θεμελιώδη μας πολιτική που είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. Η πρωτοβουλία για τους νέους φυσικά και πρέπει να υποστηριχθεί, αλλά πρόκειται για 6 δις ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της τάξης των 80 δισεκατομμυρίων. Καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την απασχόληση των νέων. Δεύτερον, Πολύ σωστά, στην ανάλυση σας αναφερθήκατε στους μαθητευόμενους. Και εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Οι νέοι αυτοί μαθητευόμενοι, στους οποίους προσφέρεται επιμόρφωση, εδώ δεν θα πρέπει στόχος των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων να είναι να τους δώσουμε κάποια επιμόρφωση απλώς και μόνο για να μην εντάσσονται στις στατιστικές των ανέργων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικός διότι στρεβλώνεται και η εικόνα με την οποία βλέπουμε εμείς τα πράγματα, αλλά βέβαια και το θέμα της αποκατάστασης των νέων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι δυνατόν να παρετηθείτε μπροστά στο Συμβούλιο. Αυτό πρέπει να το υποστηρίξετε πάση θυσία. Και εκεί θα κρυθούμε. Και θα κάνουμε ό,τι πρέπει ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες μας να γνωρίζουν ποια είναι η πραγματικότητα της πολιτικής δράσης των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό ήταν το δεύτερο. Και έρχομαι στο τρίτο. Σωστά είπατε ότι στόχος μας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων και κυρίως των νέων. Και εδώ λοιπόν πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικός όσον αφορά τη μεθοδολογία. Πώς δηλαδή, με ποια μέθοδο θα αποκατασταθούν επαγγελματικά οι πρόσφυγες. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια κατακαιρματισμένη μέθοδο. Ασχολούμαστε με τα χαρτιά, με τα διπλώματα, με τις γλώσσες. Νομίζω ότι με τον κατακαιρματισμό αυτό, πρώτο στάδιο, δεύτερο στάδιο, τρίτο στάδιο κτλ. δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη, το ζήτημα επίγει πολύ περισσότερο και έτσι το πρόβλημα της πρέπει να το πάρουμε στα χέρια μας αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν υπάρχει γλωσσική ένταξη των ανθρώπων αυτών υπάρξει επαγγελματική τους αποκατάσταση. Άρα λοιπόν, η ισοτιμία των διπλωμάτων, η επιμόρφωσή τους πρέπει, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Και πρέπει να δείξουμε τα δόντια μας στο Συμβούλιο, στους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά δεν βλέπω να επενδύουν στην πραγματικότητα της δράσης. Εμείς δεν θέλουμε λόγια. Εμείς είμαστε πολιτικοί, το ξέρετε κι εσείς πρόεδρε, ότι εδώ στην Επιτροπή μας πιστεύουμε στα έργα, όχι στα λόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το σχέδιο γνωμοδότησής σας. Περιλαμβάνει σημεία με τα οποία συμφωνούμε. Και θέλω να υπογραμμίσω κάτι για το σημείο 1, το οποίο λέει ότι το 2017. Ε, Ο προπολογισμό πρέπει να είναι στοιχείο κλειδί για να ενισχυθεί η συνεισφορά της Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και την ε, εξάλληψη της φτώχεια. Αυτό δεν πρέπει να είναι λόγια, πρέπει να είναι κάτι το οποίο όντω να ισχύσει. Επ' αυτού λοιπόν θα ήθελα και πάλι να υπογραμμίσω πόσο μεγάλη σημασία έχουν ε, τα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου για να μπορέσει να εφαρμόσει ότι πρέπει να εφαρμόσει στον προβλησμό του 2017. Χρειάζονται οι απαραίτητοι πόροι για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, φτώχειας, της παιδικής φτώχειας. Και σίγουρα Χρειάζεται δέσμευση από μας και κονδύλια, υποχρεώσεις δηλαδή, για την εγγύηση όσον αφορά την νεολαία. Το είπε και η κυρία Σαρτιά αυτό. Και έτσι έρχομαι στην απόφαση του Κοινοβουλίου του Μαρτίου, όπου στο σημείο 12 λέμε ότι όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας πρέπει να έχουν καλά προσόντα, δεξιοτεχνίες και ότι αυτά είναι προσόντα τα οποία πρέπει να προσφέρουμε και στους νέους πρόσφυγες. Αυτό σημαίνει πόρους όμως, λεφτά και επαρκή κονδύλια και για τις υπηρεσίες απασχόλησης και για το έργο τους και για το προσωπικό τους γιατί μπορούν να βοηθήσουν πολύ σε θέματα απασχόλησης αλλά και κοινωνικά. Τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γενικότερο περιθώριο των δημοσιονομικών μας προοπτικών των πολιτών για την περίοδο 2016 με 2020. Εκεί μέσα είναι και το 2017. Πόροι λοιπόν για την ανάπτυξη και την απασχόληση και κυρίως για να ανταπεξέλθουμε στους στόχους μας για την ανεργία των νέων. Και θέλω να προσθέσω κάτι. Ακούσαμε τον κύριο Γκάρτ να λέει ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστικοί. Ακούσαμε και την κυρία Χάρκιν νωρίτερα που είπε ότι δεν είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε με σαφήνεια το ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με business as usual. Ναι, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι και πέρυσι και φέτος τροποποιούμε τον προϋπολογισμό. Υπάρχει τρόπος να εκτιμήσουμε καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες και να φτάσουμε σε ένα σημείο που να αλλάζουμε τις διαδικασίες. Και μετά την πρακτική αυτή με τα trust funds, για την οποία δεν είμαι και πολύ ξεκάθαρος, το Συμβούλιο για δικούς τους λόγους το ήθελε, όλη η δημοσιονομική διαδικασία έτσι γίνεται πιο αυθαίρετη υποβάλλεται όλο και λιγότερο στο δημοκρατικό έλεγχο και κυρίως δεν εξυπηρετεί τις προτεραιότητες εκείνες τις οποίες θέλουμε να εξυπηρετεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Από το ECR η έφυγε. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Χάρκιν. Thank you. Ευχαριστώ. Στην γενική συζήτηση σήμερα ε, καταδείξαμε ποια είναι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι κι αλλά έχω και δύο. Ιδιαίτερα όσον αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση, έχουμε την εγγύηση για την νεολαία. Και ένα από τα πρώτα θέματα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι συμφωνώ με την κυρία Μόρτεν Σαρτιέ ότι ο, το Συμβούλιο χρησιμοποιεί το μηχανισμό αυτόν απλώς για να βγάζει τους ανθρώπους αυτούς από τις στατιστικές για την ανεργία. Γι' αυτό τους επιμορφώνει. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος βέβαια της εγγύησης για την ολέα. Επίσης, γίνονται και καλές προσφορές. Αν δούμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, το έχουν θέσει το ζήτημα της ποιότητας που προσφέρεται. Και δεν ξέρω σε άλλες χώρες μέλη, αλλά ξέρω από τη δικιά μου χώρα ότι γίνονται πολλές συζητήσεις για το τι είδους προσφορές γίνονται στους νέους. Και σίγουρα πολλές από αυτές τις προσφορές καθ' άλλο παρά ποιότητας είναι. Και γι' αυτό που είπατε και εσείς για την μαθητεία. Ρωτάω λοιπόν, γιατί οι νέοι πιστεύουν ότι δεν είναι δουλειά αυτό, θεωρούν ότι δεν είναι κάτι ελκυστικό. Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα. Έπειτα πολλές φορές στην Επιτροπή μας εδώ, το ξέρω, ότι έχουμε συζητήσει για το μοντέλο που στη Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες χρησιμοποιείται πάρα πολύ και ότι θα έπρεπε να το αντιγράψουν και άλλες. Προσοχή όμως, οι χώρες μέλη έχουν διαφορετικά συστήματα. Πάντως, σε μια γενική αρχή τη στηρίζω. Και όταν μιλάμε για τους νέους, οι ανάγκες του EGF και ό,τι συζητήσεις είχα εγώ τον τελευταίο καιρό δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τις ε, ανάγκες που καλύπτει το Ταμείο αυτό για τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση. Ένα από τα ζητήματα εδώ που τίθενται και που διαπιστώσαμε σε κάποιες αιτήσει που φτάνουν είναι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρχουν αρκετοί νέοι που εμπλέκονται για, ως δικαιούχοι του ταμείου αυτού. Άρα και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο αυτό όσο γίνεται περισσότερο επίσης χρησιμοποιείται για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μου, για το Άλντε. Όπως επίσης και η δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Σήμερα, 9 με μισή ήμουν σε μια από τις πιο καταπληκτικές συναντήσεις τις οποίες έχω πάει ποτέ για την ψηφιοποίηση και γενικά για τις ε, τραπεζικές υπηρεσίες, ε, πληρωμές και άλλα. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες. Και σκέφτομαι και εγώ τώρα και προσπαθώ να βάλω μια τάξη στο μυαλό μου για το πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά όταν μιλάμε για απασχόληση. Κάτι που δεν πρέπει να γνωρίζει βέβαια και ο προπολογισμό μας. Και τέλος το θέμα της φτώχεια των παιδιών, στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί μέχρι τώρα. Ναι, οι γονεί πρέπει να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά για να μπορούν να βοηθήσουν να μην υπάρχει αυτή η φτώχεια των παιδιών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες για μένα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίνων δεν έχω εδώ κανέναν, ούτε για το EFTT. EFN. Παρακαλώ, κύριο Μάτο. Ευχαριστώ, εισήγητα. Είναι λογικό, μιας και είμαστε η Επιτροπή για τα κοινωνικά θέματα, να βρίσκουμε τα στοιχεία που περιλαμβάνεται στο πρώτο τμήμα, ότι πρέπει να βοηθήσει δηλαδή τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το δύο είναι η στόχευσή μας στην ανεργία των νέων, είναι βασική μας ανησυχία. Κάποια στιγμή σε μια επιτροπή είχαμε δει ότι οι νέοι από 16 μέχρι 25 ε, μέχρι τα 30 πήγαμε μετά και τώρα ξαφνικά πάμε τους νέους μέχρι και τα 40. Και όλους αυτούς θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να μπουν στην, στον κόσμο της εργασίας γιατί η φιλανθρωπική βοήθεια η οποία χορηγείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι λύση. για το σημείο 3, για τις λιγότερο ευνοημένες κατηγορίες του πληθυσμού όπως ε, ε, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι μειονότητες. Τώρα τι θα πει αυτό μειονότητες, ε, πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο. Το σημείο 4. Κάποια προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το σημείο 5 επαγγελματική κατάρτιση, συνεχής κατάρτιση διαβίου κατάρτιση. Πρέπει να προσέξουμε γιατί μέσα από αυτά τα συστήματα κατάρτισης μερικές φορές αποκρύβουμε, καλύπτουμε τους αριθμούς τους, της ανεργίας. Είναι της μόδας. ψηφιγοποίηση προφανώς πολύ σημαντικό, το 7. Προώθηση της επιχειρηματικότητας. Το 8 κοινωνικά θέματα, θέματα προστασίας των εργαζομένων, για το σύνολο των χωρών της Ένωσης, γιατί δυστυχώς οι διαφορές μεταξύ τους είναι τεράστιες. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και με εκπλήσει λίγο, ότι δεν αναφέρεστε καθόλου στις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες κατά 90% εποφελούνται από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παγκοσμιοποίηση. Αυτό το οποίο με εκπλήσει λιγότερο και το είχα πει και προφορικά. Ναι, στις μικρομεσαίες, αλλά πώς. Σε καμία περίπτωση στα εννέα σημεία τα οποία περιλαμβάνετε δεν αναφέρεστε στη συγκεκριμένη βοήθεια. Μιλάτε εσείς όταν μιλάτε προφορικά αλλά δεν το γράφετε. Και στο σημείο 9. Εδώ είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος εκφράζεται ελπίδες, ελπίδες φρούδες ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να βοηθήσει την ολοκλήρωση της ενίας αγοράς. Εμείς είμαστε κατά φυσικά γιατί δεν λειτουργεί. Μιλάτε για ανταγωνισμό και για κοινωνική σύγκλωση. Πού τα είδατε αυτά. Α, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Πού το είδατε. Και επίσης εφαρμογή των κοινωνικών προτύπων. Ε, καλά κάνετε και το ζητάτε αυτό, αλλά εδώ και δεκαετίες εμείς διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν γίνεται, δεν λειτουργεί το σύστημα. Μάλιστα. Κάποιες ερωτήσεις από τη συζήτηση. Καταρχάς, ε, πρόκειται για μια εντολή για τριμερή διάλογο, όχι για ένα ευρύ ε, έγγραφο εργασία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το θέμα τη ε, γενικότερη ανεργία των νέων και τη αντιμετώπιση του. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να τονίσω ότι μιλάμε για το θέμα της υποστήριξης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τουλάχιστον στη Γερμανία. Αυτό έχει να κάνει με το 70% των θέσεων κατάρτισης. Και στη Γερμανία έχουμε 140.000 τέτοιες θέσεις κατάρτισης που δεν έχουν πληρωθεί, που δεν έχουν ε, δοθεί σε κάποιον και συχνά στη Γερμανία ακούμε ότι θα ήθελε κάποιος ε, να δώσει τη θέση αυτή κατάρτιση σε κάποιον ε, νεαρό μετανάστη που έχει δύο τραυματικέ εμπειρίε, αλλά δεν υπάρχει ειδικό κόσμο με ειδική κατάρτιση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Και γι' αυτό λοιπόν στο σημείο αυτό λέμε ότι μπορούμε να δώσουμε πόρου προκειμένου να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις που θα φρόντιζαν για την κατάρτιση και εκπαίδευση των νεαρών προσφύγων. Αυτό εννοούσα την πρακτική υποστήριξη, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να διευκρινιστεί στην διαπραγμάτευση, στο πεδίο εντολή, θα πρέπει να τύχει διαπραγμάτευση καταρχά. Και κατά δεύτερον θα πρέπει να αποτελέσει ένα ποιοτικό πρόγραμμα, το οποίο στην επόμενη φάση των εργασιών της Επιτροπής μας ε, θα πρέπει να τεθεί στα πλαίσια της επεξεργασίας του προϋπολογισμού και αν το καταθέσουμε ως πρόταση από όλες τις ομάδες, νομίζω ότι θα υπάρχουν αντιθέσεις από οποιαδήποτε πλευρά και θα πρέπει να κοιτάξουμε το κείμενο που θα τυπωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα της πρόθεσης αυτής. Αυτά σε ό,τι αφορά τα πολιτικά προγράμματα και το προπολογισμό. Τρίτο σημείο, σε ό,τι αφορά αυτό που σχολιάστηκε για τις θέσεις μαθητείας. Οι θέσεις μαθητείας θεωρώ ότι είναι πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξεύρεση του σωστού επαγγέλματος ή για τη συμπλήρωση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν υποκαθιστά όμω αυτό τίποτα, γιατί συχνά ε, το θέμα στη Γερμανία της ε, κατάχρησης των θέσεων μαθητείας ε, με μηδενική αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ο στόχος αυτός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός μας να κάνει τρεις-τέσσερις τέτοιες θέσεις μαθητείας ο νέος ε, χωρίς να πληρώνεται. Πρόκειται για μια καταχρηστική πρακτική. Αυτή η πρακτική λοιπόν η καταχρηστική υπάρχει και άρα δεν επικεντρώνομαι στο θέμα της μαθητείας. Το θέμα είναι η σωστή ουσιώδης και καλή σωστή ε, εκπαίδευση η επαγγελματική, είτε μέσω πανεπιστημίων και τεχνικών σχολών, είτε μέσω μαθητείας. Και η κατάχρηση τέτοιων ε, πρακτικών είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να θα απασχολήσει. Αυτά για τη ε, συζήτηση αυτή. Πρόθεσμη για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 11η Μαΐου. 15 Μαΐου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού στις 13 Ιουνίου. Και να σας καλέσω λοιπόν, αν θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες για την ε, τροποποίηση της εντολής. Και περνάμε λοιπόν στο σημείο 6 της ε, ημερήσιας διάταξης. Έχουμε καθυστερήσει σημαντικά σήμερα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το λόγο έχει ο Τζορς να είναι σύντομο, να είσαι σύντομος, ε, Τζορτ. Ευχαριστώ, αξιότιμε πρόεδρε και συνάδελφοι. Νομίζω ότι χρειάζεται. Ο, θεωρώ να σα δώσω ιδιαίτερα το υπόβαθρο τη ε, πρόταση αυτή. Το 2008 ψηφίστηκε η οδηγία για τι εκδομικέ Υπηρεσίε και κλείθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τέσσερα χρόνια να μας υποβάλει μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας. Πρόκειται για ένα κλάδο ο οποίος βρίσκεται σε μια φάση μεταμόρφωσης. Τεχνολογικές, ε, τεχνολογικοί παράγοντες, τεχνολογικές εξελίξεις. Και πιστεύω ότι αυτός ο τομέας αφενός μέσω των καθολικών υπηρεσιών αλλά αφετέρου και μέσω των ταχυδρομικών υπηρεσιών περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικούς τομείς. Άρα δύο τομείς ε, ουσιαστικά συνενώνται σε έναν. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρχάς διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ε, επαρκή αξιόπιστα στοιχεία και αυτό συχνά μας αναφέρεται ότι είτε είναι παροχημένα τα στοιχεία που δίδονται του 2012 για παράδειγμα, είτε ότι δεν τα, δεν τα διαθέτουν τα κράτη-μέλη οι, οι εκάστοτε κλάδοι τα στοιχεία αυτά τα απαραίτητα. Άρα υπάρχει μια έλλειψη επαρκών αξιόπιστων, στοιχείων. Ένα άλλο θέμα. Τα προϊόντα των υπηρεσιών των διάφορων παρόχων είναι πολύ ε, παρόμοια και μπλέκονται και αυτό μας δυσκολεύει σε θέματα διαφάνειας. Και γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι η εντολή μας είναι να υποδείξουμε στους υπαλλήλους, στους απασχολούμενους του κλάδου αυτού, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας. Το 2013 είχαμε περίπου 2 εκατομμύρια απασχολούμενους στον τομέα αυτό. αλλά σε ό,τι αφορά τα πακέτα express δεν μπορούμε παρά να κάνουμε εικασίες, 270.000 για παράδειγμα και σε ό,τι αφορά το 2010. Σε ό,τι αφορά τους απασχολούμενους στον τομέα των καθολικών υπηρεσιών, πρέπει να σας πω ότι ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε κατά 4% κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει ότι καλωσορίζουμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων που προσπάθησαν από κοινού με τους απασχολούμενους ε, στον τομέα αυτό να διασφαλίσουν τους όρους εργασίας στον κλάδο αυτό. Δεν είναι φυσικά οι καλύτερες δυνατές ε, συνθήκες αυτές, αλλά παρά όλα αυτά ε, υπήρξαν κοινωνικές ε, συμβάσεις, συλλογικές κοινωνικές συμβάσεις για την μεταβατική αυτή φάση στον κλάδο αυτό και όπως σα είπα υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ των παρόχων καθολικών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Έχουμε και προβλήματα με τους ψεταπασχολούμενους και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να επικρίνουμε τις ε, επισφαλείς και ευέλικτες ε, συμβάσεις εργασίας στον τομέα αυτό και επειδή στην πράξη ναι μεν τηρούνται τα επίπεδα μισθών αλλά οι όροι εργασίας οδηγούν σε μεγάλο άγχος σε πολλές υπερορίες και αυτό στο μέλλον θα αυξάνεται και θα πηγαίνει πολύ φοβόμαστε αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ένα τελευταίο σημείο, επιτρέψτε μου να επισημάνω, το οποίο, μάλλον πρώτο τελευταίο σημείο που θέλω να επισημάνω, είναι η σημασία τη ε, ε Αυτό πήγε αρκετά καλά στον κλάδο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, είναι μεγάλη μεταβατική φάση που περνάει ο κλάδο αυτό και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι η μετεκπαίδευση, η αλλαγή ε, εκπαίδευση και η συμμετοχή σε κοινωνικέ επιτροπέ. Χρειαζόμαστε επιπλέον ε, στοιχεία και καλωσορίζουμε και την ε, Επιτροπή για τον Τομιακό Διάλογο σε ό,τι αφορά τις εγκεντρωμικές υπηρεσίες. Ε, γνωρίζετε τα προβλήματα που είχαμε και σε ό,τι αφορά την κατάρτιση της έκθεσης. Εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, προσβλέπω και στη συνεργασία με τους κοιόδες εισηγητές και φυσικά στα δικά σας σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και η επόμενη είναι η κυρία Στάινρουκ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Ζορμπαχ. Μπαχ. Σας ευχαριστούμε για την καλή γνωμοδότηση και για τις καλές Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω, γιατί όλες οι πτυχές που έχουν σημασία για το ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν καλυφθεί. Παρ' όλα αυτά θα καταθέσω και εγώ κάποιες τροπολογίες από πλευρά της ομάδας μου σε ό,τι αφορά τις αλυσίδες υπεργολαβίας που στον τομέα αυτό διαμορφώνονται με πολύ δύσκολο τρόπο σε ό,τι αφορά και το ωράριο εργασία, σε ό,τι αφορά την τήρηση των όρων ανάπαυσης. Θέλουμε πιο πολλούς ελέγχους εργασίας και σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να υπάρχει τρίτη δραστηριοποίηση. Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές εξελίξεις τώρα, μιλάμε για την ψηφιοποίηση, για την εξέλιξη των μέσων. και πώς μπορούν οι πάροχοι και οι προμηθευτές να χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους. και κατά πόσον επηρεάζεται και η εκπαίδευση των εργασιών από τις ε, νέες τεχνολογικές ε, ε, εξελίξεις. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λοτόφσκι τώρα από το ECR. E, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρότασή σας, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να σχολιάσει κανείς. Τι εννοώ. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία νομίζω έχουν πολύ μεγάλο βάρος. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στον τομέα των ταχυδρομικών οι εργαζόμενοι παίζουν έναν κρισιμότατο ρόλο, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι κάνουν τη σκληρή θα έλεγε κανείς δουλειά. Στον ταχυδρομικό τομέα δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το θέμα δεν είναι αμοιβέ. Το θέμα είναι η σταθερότητα των θέσεων απασχόλησης, η κατάρτιση η σωστή και η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στα πλαίσια της ψηφιοποίησης. Πολλές φορές η επιχείρηση ταχυδρομική ανήκει στο κράτος, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση τα κράτη είναι αυτά τα οποία έχουν την ευθύνη να βελτιώσουν τα επίπεδα και να αντιμετωπίσουν ε, προβληματικές μορφές απασχόλησης που δεν επιτρέπουν στους εργαζομένους να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα μέσα. Ο ανταγωνισμός στον ταχυδρομικό τομέα δεν οδηγεί σε βελτίωση στις συνθήκες εργασίας, αλλά οδηγεί σε ε, θύματα στον τομέα των τιμών και των ε, πελατών. Οι εταιρείε κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν τους διαγωνισμούς και αυτό οδηγεί σε μια πτώση της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών και σε υπερβολές σε σχέση με το σεβασμό των κανόνων εργασίας. Στην Πολωνία, σαν παράδειγμα, είχαμε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία εργαζόταν εξ ονόματος του, ε, μάλλον και για το κράτος, εργολαβικά, ήταν ε, φυσικά πολύ φθηνή η εταιρεία αυτή, αλλά οι συνθήκες εργασίας ήταν εφικτές. Ο ανταγωνισμός σε μια οικονομία φυσικά και έχει μεγάλη σημασία, αλλά οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους. Ο ταχυδρομικός τομέας είναι στρατηγικός τομέας για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το κράτος. Γι' αυτό λοιπόν τα δικαιώματα των εργαζομένων ταχυδρομικών θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρκινγκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι μια συζήτηση η οποία κρατάει εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε συζητήσει επανειλημμένα τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών των ταχυδρομικών και οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2010 δεν επιτρέπουν να καταλήξουμε ε, στο τι πραγματικά συμβαίνει. Οι αλλαγές είναι συνεχείς και τα αποτελέσματα είναι αμφίβολα. Ε, ο τομέας αυτός μειώνεται 4 περίπου τις 100 από χρόνο σε χρόνο, ο κύκλος εργασιών του εννοώ, και σε ορισμένες χώρες μέλη οι αρχές επί του προϋπολογισμού έχουν καταδικάσει τις υπηρεσίες που ασχολούνται με, την ε, ταχυδρομική, ε, με τις ταχυδρομικές δραστηριότητες διότι λειτουργούν μέσα σε καθεστώτα ολιγοπολίων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτό το οποίο μας απασχολεί εδώ βέβαια είναι η απασχόληση και οι συνέπειες της εργασίας στις συνθήκες ε, κάτω από τις οποίες διεξάγεται. Ε, εγώ δεν έχω προχωρήσει σε βάθος, αλλά παρόλα αυτά οι παροχές υπηρεσιών στον τομέα αυτό συνήθως παρέχουν συνθήκες εργασίας επαρκής ε, στα πλαίσια συλλογικών συμβάσεων και σωστή κοινωνική διαχείριση των νέων μέσων εργασίας, ιδιαίτερα της ψηφιοποίησης πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση από κοντά στη δική μου χώρα, στην Ιρλανδία, και εδώ θυμίζω ότι κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ένα από τα θέματα τα οποία μας ανησυχούν είναι το θέμα του κλεισίματος των ταχυδρομικών γραφείων της Υπέθρο. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό συνδέεται με αυτά που συζητάμε, αλλά για τις γεωργικές περιοχές αυτό είναι ένα πρόβλημα. και το κλείσιμο αυτών των γραφείων που έκαναν ταυτόχρονα πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες είναι ένα χτύπημα για τις περιφέρειες. Πάντως, ευχαριστώ για το έγγραφο, δεν μπορώ να προσθέσω πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και μην δεν τον βλέπω. Υπάρχει κάποιος άλλος εκπρόσωπος σε ομάδας Καρίμα Ντελή, ούτε αυτή τη βλέπω από τους πράσινους, κάποιος άλλος να την αντικαθιστά. Όχι. Λάουρα Ετζέα. Τη Λάουρα τη βλέπω. E ah, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα, λέει η κυρία Τζέα, να ευχαριστήσω τον κύριο Μπακ, με τον οποίο θα συνεργαστούμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο προσπάθησα να κάνω είναι να αναζητήσω την διαδικασία της οδηγίας αυτής και ποιο είναι το στάδιο της εφαρμογής στις διάφορες χώρες και κυρίως στη δική μου χώρα για να καταλάβω πώς έχει το παζλ αυτό. Το κοινοτικό πλαίσιο των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων καλύπτεται από μία πρώτη οδηγία του 77 που προχώρησε σε μία αρχή της διαδικασίας απελευθέρωσης. Μετά υπήρξε μία μεταρρύθμιση η οποία θεωρητικά οδήγησε στο πλήρες άνοιγμα της αγοράς το 2010 για τις περισσότερες χώρες όπως και τη δική μου. Από την 1η Ιανουαρίου του 2011 λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχουν αποκλειστικά δικαιώματα για μία επιχείρηση κρατική. Σύμφωνα με το άρθρο 1 λοιπόν της οδηγίας η Ιταλική κυβέρνηση έχει καταργήσει πλέον το μονοπόλιο το οποίο ίσχυε μέχρι το τέλος του 10 υπέρ της εταιρείας Poste Italiane. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια οδηγία ακριβώς για την απελευθέρωση, κάτι το οποίο όμως επέτρεψε να δοθεί στην Poste Italiane η λειτουργία των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων για 15 χρόνια με επαλήθευση της διαδικασίας και των συνθήκων ανά 5 χρόνια. Σπάσαμε το μονοπόλιο, αλλά στην ουσία δώσαμε τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών στο ίδιο το μονοπόλιο. Από τη μία λοιπόν η Ιταλία λέει ότι θα φιλελευθερωποιήσει τις ταχυδρομικές δραστηριότητες, στην ουσία όμως άφησε τα πράγματα ως έχουν και εξακολουθεί να δώσει μια λοιπον η ιταλια λεει οτι θα φιλελευθεροποιήσει τις ταχυδρομικες κυρίαρχη θέση στα Ιταλικά ταχυδρομεία, την Poste ιταλιανη που ανήκει και στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων της χώρας και στο Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών κτλ. Θα δούμε λοιπόν πώς εννοούν στο μέλλον να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μπήκαν στην αγορά, αλλά από ό,τι φαίνεται η αγορά αυτή μέχρι τώρα δεν είναι πραγματικά ανταγωνιστική και δεν γίνονται σεβαστά τα κριτήρια της κοινοτική οδηγίας. Έχουμε απελευθερώσει την αγορά αφήνοντας όμως το μονοπόλιο ε, στην ίδια εταιρεία που ήταν ιδιοκτήτη στο παρελθόν. Έτσι έχουν τα πράγματα στην Ιταλία, θα κάνουμε τις αξιολογήσεις μας και υπό το φως των συμπερασμάτων θα συνεργαστούμε με τον κύριο Μπάκ. Mara Eh, Σύντομα, το στάδιο εφαρμογής της οδηγίας στην Ιταλία δεν υπάρχει ουσιαστικά από πλευράς των καταναλωτών. Όπως είπε και η συνάδελφος, η Πόστε Ιταλιάνε έχει το μονοπόλιο των ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν κάνει αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει, να παραδίδει τα γράμματα. Έχει γίνει τράπεζα, έχει γίνει μια εταιρεία, μια επιχείρηση πουλάει τα πάντα από στυλό μέχρι παιχνίδια και σύν τη άλλη η Ιταλιάνε είναι και ένας από τους σημαντικούς μετόχους της Αλιτάλια. Δηλαδή έγινε μια μεγάλη επιχείρηση, κάτι το οποίο δεν είναι αρμοδιότητα. Αυτό που δεν κάνει είναι να παραδίδει γράμματα. Ακόμα και στη δική μου εκλογική περιφέρεια, εγώ κατοικώ σε μια παιδινή περιοχή, αλλά έχουμε δυσκολίες. Τα γράμματα φτάνουν μία φορά τη βδομάδα. Σκεφτείτε τι γίνεται στις ορεινές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό ε, και αν υπάρχουν καθυστερήσεις, επληρωμές και τα λοιπά υπάρχει επιβάρυνση για τους πολίτες. Το θέμα είναι σοβαρό και γι' αυτό πάρα πολλοί δήμαρχοι έχουν στείλει επιστολές όχι μόνο στο Υπουργείο αλλά και σε άλλες αρχές ζητώντας παρεμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει τον τρόπο που λειτουργεί η εταιρεία αυτή, όπως και ελέγχει την είσοδο της Πόστε Ιταλιάνε στην Αλιτάλια γιατί δεν φέρει εις πέρα στις ανηλυμένες της υποχρεώσεις. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται είναι μια χρήσιμη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξει την εφαρμογή ε, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Ιταλία που δεν γίνεται σωστά. Καλώς περνάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Χάουιτ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τη συνάδελφο Στάνμπρουκ και συμφωνώ με αυτά που είπε. Ο κύριος Μπαχ μας έδωσε μια πολύ καλή παρουσίαση και πολύ καλά τα είπε. Το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις καθολικές υπηρεσίες. Στηρίζω λοιπόν τους κοινωνικούς εταίρους ε, στην προσπάθεια συνεργασίας. Όσον αφορά λοιπόν τις καθολικές υπηρεσίες, 89% του κόσμου στη χώρα μας, στον Ηνωμένο Βασίλειο, τις υποστηρίζουν. Και είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε και πάλι την υποστήριξή μας στις υπηρεσίες αυτές αν στο τέλος συζήτηση θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαντικό είναι να μας πούν ποια είναι δικιά τους η θέση για τις καθολικές υπηρεσίες και τις επιπτώσεις στην απασχόληση. του, είπε και ο κύριος Ζομπάχ σήμερα. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει να πει γι' αυτό. Τώρα κάτι που δεν αναφέρθηκε είναι το πώς οι καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες υπονομεύονται από cherry picking, δηλαδή από επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται, παίρνουν ένα κομματάκι το οποίο τους εξυπηρετεί γιατί τους κάνει να κερδίζουν πολλά και έτσι υπονομεύονται οι καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Δεν ξέρω ο κύριος Μπάχ τι έχει να πει γι' αυτό, ποια είναι η γνώμη του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να το σχολιάσει κυρίως μάλιστα μετά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την διασυνοριακή μεταφορά δεμάτων. σε σχέση με το status quo και με τη διατήρηση των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών. Κάποιοι από αυτούς τους φορείς που έρχονται και παίρνουν τα κομματάκια εκείνα που τους αποδίδουν περισσότερα καταστρέφει ακόμα περισσότερο γιατί αν μη τι άλλο δεν επιτρέπει στις ταχυδρομικές υπηρεσίες να παίζουν επίσης ώρες το παιχνίδι. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Μπαχ να πει τη γνώμη του γι' αυτό. Οι σοσιαλιστές μάλλον θα υποβάλουμε κάποια τροπολογία για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Κρίστοφερ Φίτμαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παχ για την εξαιρετική του έκθεση. Γνωμοδότηση, πιο σωστά. Δύσκολα θα διαφωνούσε κανείς με αυτά τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή. Πάντως, επιτρέψτε μου με κάθε ταπεινότητα να ζητήσω κάτι από τον κύριο Παχ. Ίσως θα μπορούσε να είναι πιο απόλυτο στις συστάσεις του, κυρίως όσον αφορά ε, τους ανθρώπους που απασχολούνται στον κλάδο αυτό. Πολλά λέμε για την απορρίθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ότι υπάρχουν ωφέλη από αυτήν, αλλά επίσης, δυστυχώς, υπάρχουν και κακές συνέπειες. Η κυρία Χάρκιν το ανέφερε, είπε ότι σε μικρές πόλεις, σε χωριά, τα ταχυδρομικά γραφεία και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες εξαφανίζονται. Και δεν είναι μόνο αυτό είναι επιπλέον ότι ο ανταγωνισμός συμβαίνει σε βάρος των εργαζόμενων. Γιατί οι εμπορικές επιχειρήσεις θέλουν να μειώσουν το κόστος και από πού κόβουν κόστος εισάγουν ευέλικτες μορφές εργασίας κάτι το οποίο είναι πολύ κακανέα για τους εργαζόμενους. Ο κύριος Μπάχ λοιπόν κάνει κάποιες πολύ καλές συστάσεις, αλλά τον παρακαλώ να τις ε, διατυπώσει με πιο έντονο τρόπο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Φαντούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχοντας εργαστεί επί 30 χρόνια στα ελληνικά ταχυδρομεία, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ένας κλάδος που σιγά σιγά σβήνει. Το αντικείμενο του ταχυδρομείου, η επιστολή, έχει στην κυριολεξία εξαφανιστεί. Ποιο στέλνει σήμερα γράμματα, επιστολές. Όλοι επικοινωνούμε με τα email και με άλλου τρόπου. Το πολύ πολύ να στείλουμε κάποια ευχητήρια κάρτα τα Χριστούγεννα ή το, το Πάσχα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να κοιτάξουμε σαν Επιτροπή απασχοληση είναι η μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότηση στα ταχυδρομεία δεν αναπληρώνεται. Αυτό γίνεται πρώτον γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας αρκετό, αλλά προσπαθούν να μειώσουν και το λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα να πιέζουν οι εργαζόμενοι να αναπληρώσουν το κενό. Εγώ πήγα μια επίσκεψη στο ταχυδρομείο που εργαζόμουν, ήταν 8 άτομα εκεί παλιά και τώρα 2 άτομα καλούνται να βγάλουν όλη τη δουλειά σε απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις έχουν καταργηθεί, δεν γίνονται συλλογικές συμβάσεις εργασία και δεν, γίνεται, δεν σέβονται οι επιχειρήσεις στην δικιά μας περίπτωση, τα ελληνικά ταχυδρομεία, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν μπορούν να πάρουν άδεια, ε, δουλεύουν ενώ είναι άρρωστοι, δεν μπορούν να λείψουν από την υπηρεσία τους. Ε, το δίκτυο των ταχυδρομείων είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να στραφούν για να αναπληρώσει το κενό σε νέες υπηρεσίες. Γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το δίκαιο. Αλλά οι συλλογικές συμβάσεις οι οποίες δεν εφαρμόζονται έχουν δώσει χώρο σε κάποιες εταιρείες οι οποίοι νοικιάζουν εργαζόμενους στα ελληνικά ταχυδρομεία. Το κόστος δεν είναι μικρότερο για τα ελληνικά ταχυδρομεία, αλλά οι αμοιβέ και οι συνθήκε εργασία των εργαζομένων είναι πολύ κατώτερε από αυτέ που πρέπει. Επίση, αναφέρθηκαν συνάλφοι για το κλείσιμο των ταχυδρομικών γραφείων τη επαρχία, τα οποία ήταν πολύτιμα για του ανθρώπου που κατοικούν σε απομακρυσμένε περιοχέ. Βέβαια τα ταχυδρομεία έχουν στραφεί σε άλλε μορφέ τώρα, έχουν γίνει τράπεζε, εξοφλήσει λογαριασμών κτλ. Ε, επί τη ουσία, συμφωνώ με πάρα πολλά από τη, στην έκθεση, απλώς θα έπρεπε να γίνεται αν και δεν το θέλουμε αυτό, περισσότερος έλεγχος αν εφαρμόζονται αυτά που πρέπει να εφαρμοστούν για την προστασία των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και έτσι ολοκληρώθηκε ο κύριος των ομιλητών και πρώτα δώσω το λόγο πάλι στον εισηγητή τον κύριο Μπαχ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι την επόμενη φορά όταν σας ε, φέρουν ε, ένα ταχυδρομικό πακέτο θα πρέπει να μιλήσετε με τον διανομέα σας, ε, με τον ταχυδρόμο, για τις ε, συνθήκες εργασίες του. Γιατί μας λένε ότι σε πολλές περιπτώσεις πολλά πρέπει να ρυθμίσουμε. Υπάρχει ένας ελάχιστος κατάδοτος μισθός και αυτό παίρνουν τα ταχυδρόμοι. Αλλά στις 8 ώρες που ε, πληρώνονται, για τις οποίες πληρώνονται, έχουν τόσο πολλά πακέτα και γράμματα να δώσουν που δεν τους φτάνουν οι 8 ώρες. Χρειάζονται 10 και 12 και σε κάποιες περιπτώσεις. Εδώ ε, ε, μιλάμε λοιπόν για κατάχρηση και όχι μόνο στη Γερμανία φαντάζομαι, αλλά και σε άλλες χώρες. Και σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε θέση προς αυτό στην έκθεση αυτή και σας παρακαλούμε να μας υποστηρίξετε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπάχ για να κλείσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι το δέχομαι απόλυτα αυτό το επιχείρημα και σίγουρα από πλευράς και των άλλων συναδέλφων θα ακούσουμε τι γίνεται και θα ενισχύσουμε φυσικά τις συστάσεις μας στην έκθεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα μια γενική ε, παρατηρήση, καταρχά να πω ότι χαίρομαι για την γενικότερη υποστήριξή σα, αλλά μια γενική διαπίστωση να κάνω καταρχά. Είναι μια γνωμοδότηση αυτή. Μια έκθεση προ την. Ε, σε ό,τι αφορά τι κοινωνικέ μορφέ απασχόληση, ε, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και ο κύριος Φέρμπερερ τα τα θέματα αυτά και χαιρόμαστε λοιπόν. Και αυτό με οδηγεί στη σκέψη της κυρίας Χάρκιν, η οποία λέει ότι με την απόφαση για τις οικονομικές υπηρεσίες στην Υπετρό αναφέρθηκε αυτό και από διαφόρους άλλους συναδέλφους. Η οδηγία προδιαγράφει την τήρηση των βασικών όρων και τη διαθεσιμότητα χωρίς οποιαδήποτε διακριτική μεταχείριση και νομίζω ότι όταν μένει κανείς ε, στην Ήπεθρο ε, και κλείνουν τα γραφεία και δεν ε, υπάρχουν οι ταχυδραμικές υπηρεσίες που θα έπρεπε, αυτή η διαθεσιμότητα αποτελεί διακριτική μεταχείριση λοιπόν. Ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση και αυτό το βλέπουμε και στην έκθεση για τις οικονομικές δομές. Θα πρέπει να το δείξουμε. Διάφοροι συνάδελφοι νομίζω το ε, έδειξαν η κατάσταση στην Ιταλία κτλ. κτλ η οποία κρίνεται ε, μη ικανοποιητική και ο συνάδελφος Χάουιτ ανέφερε διάφορες επικριτές υπηρεσίες η οδηγία για τις οικονομικές υπηρεσίες προβλέπει ότι η καθολική και η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να δεσμεύει τα κράτη-μέλη για την εξασφάλιση των υπηρεσιών αυτών σε ό,τι αφορά ε, για τις πέντε εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον κτλ. Και σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό θα πρέπει να υποδείξουμε ότι οι καθολικές υπηρεσίες αποτελούν ένα μεγάλο πίτευμα του παρελθόντος και όχι μόνο για, τα, για τις αστικές περιοχές, αλλά και για την Ήλπετρο και για τις κοινωνικές εξελίξεις, τους κοινωνικούς όρους στους Δήμους και στις κοινότητες. Άρα συνολικά χαίρομαι για τη συνεργασία και το ενδιαφέρον το οποίο ε, έδειξαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό για το πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και προσβλέπω και στη μελλοντική μα συνεργασία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και έτσι περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε καθυστερήσει φρικτά, λέει ο Πρόεδρος, για την έκθεση Φέι, με πρόσφυγες στην κοινωνική δεξιότητα μέχρι την εργασία Έχουμε 45 λεπτά. Ο Μπράντο μιλάει πάρα πολύ ε, γρήγορα. Ελπίζω να τα βγάλει πέρα. Μπράντο, έχεις το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική τους δουλειά μέχρι τώρα. Οι τροπολογίες που έχουν καταθέσει περιλαμβάνουν πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία θα λάβω υπόψη στις συμβιβαστικές μου. Ποιοτικά οι τροπολογίες αυτές είναι υψηλού επίπεδου και με βοηθούν ιδιαίτερως. Ε, είμαι ευγνώμων λοιπόν. Γιατί στόχος μου είναι να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο συγκεκριμένο αλλά και να δώσουμε μία όθηση στην συζήτηση που γίνεται για το θέμα αυτό στην κοινή γνώμη. Κανένα από τα κεντρικά σημεία της πρότασής μου δεν έτυχε αντίθετης άποψης και απόρριψης όλοι εκτός από την άκρα δεξιά θεωρούν ότι η ενσωμάτωση των προσφύγων είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι κεντρικός στόχος. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και συμφωνείτε οι περισσότεροι με τα μέτρα τα οποία μπορεί να ληφθούν έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των προσφύγων στον τομέα της εργασίας, όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι ζητούν να απασχοληθούν αλλά και για τα συστήματα υγείας τα οποία σε διάφορες χώρες ε, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και τα λοιπά. Δεν υπάρχει μία συνταγή για όλους. Θα ήθελα να κάνω κάποια πιο συγκεκριμένα σχόλια σε σχέση με τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο κύριος Μαν έχουν υπογραμμίσει πολύ σημαντικά στοιχεία όπως η ανθρωπιστική κρίση και οι εξωτερικές αιτίες της κρίσης αυτής. Εδώ συμφωνούμε και σε σχέση με τα δικαιώματα των προσφύγων αλλά και τα καθήκοντά τους, τις υποχρεώσεις τους. Αυτές τις προτάσεις τις συμμερίζομαι. Σημερίζομαι επίσης και με την πρόταση οι διαδικασίες ασύλου να γίνονται σε ατομική βάση και να μην χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή για την οικονομική μετανάστευση. Αυτό θα λειτουργήσει εις βάρος αυτών που την χάνουν διεθνούς προστασίας. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από νόμιμα μέσα ε, για την οικονομική μετανάστευση, τα οποία πρέπει να είναι δίκαια και αποτελεσματικά. Ε, κάποιες ε, χώρες έχουν κάνει συγκεκριμένες προτάσεις ε, για τις χαμηλότερες αμοιβέ με τις οποίες θα πρέπει να πληρώνονται οι μετανάστες και αυτό δημιουργεί προβλήματα ξενοφοβίας και κοινωνικού ντάμπινγκ. Η αγορά εργασίας πρέπει να είναι ενιαία για όλους χωρίς διακρίσεις. Συμφωνώ επίσης και με αυτά τα οποία είπε Στίβενς ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για τον πρόσφυγα με πικεφαλαίο, αλλά κάθε άνθρωπος ο οποίος ζητά προστασία και έχει συγκεκριμένες ανάγκες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να λειτουργήσουν τα κοινωνικά ταμεία με πιο διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω ότι συμφωνούμε λοιπόν εδώ απαιτείται μια μεγαλύτερη ίσως ευελιξία της αγοράς εργασίας για την απορρόφηση των προσφύγων. Αυτό είναι λίγο θεωρητικό βέβαια και δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό σαν θέμα για την συγκεκριμένη συζήτηση. Το θέμα είναι να δούμε η ποιότητα των θέσεων εργασίας σε ποιο βαθμό βοηθά την κοινωνική συνοχή. Για τους φιλελευθέρους η κυρία Βέμπερ παρουσίασε τροπολογίες για την ενίσχυση της ταχύτητας δράσης για την ενσωμάτωση των ε, προσφύγων για να αποφευθεί ο κίνδυνος απομόνωσης. Διαρωτώ με αν θα ήταν δυνατό να υποσταριχθεί η δική μου πρόταση έτσι ώστε το κοινωνικό ταμείο να αναλάβει την βασική του δραστηριότητα, την πολιτική συνοχής ε, μέχρι το 5%. Από εκεί και πέρα αυτές οι παρεμβάσεις καθίστανται επιτακτικές λόγω του χαρακτήρα του έκτακτου των φαινομένων των μεταναστευτικών. Η πρόταση την οποία κάνετε εσείς δεν απαιτεί μια αύξηση του προϋπολογισμού αλλά μια ανακατάταξη των δαπανών στο εσωτερικό του προϋπολογισμού. Η σκιώδης εισηγήτρια της Γκουε, η κυρία Πένια, υπογράμμισε την δύσκολη κατάσταση στην οποία ζουν οι πρόσφυγες και ε, θα έλεγα υπογραμμίζει την σημασία σεβασμού των βασικών δικαιωμάτων όπως η κατοικία, η υγεία, η κοινωνική προστασία. Εδώ σημειώνεται η ανεπάρκεια των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Συμφωνώ σε αυτό. Υπογραμμίζεται η σημασία επίσης της λήψης υπόψη των επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφύγων χωρίς αυτό να επηρεάζει το αίτημά τους για χορήγηση ασύλου. Αυτό θα ήταν παράνομο σε επίπεδο διεθνούς ένομης τάξης στη σκιώδη εισηγήτρια των Πρασίνων, την κυρία Λάμπερντ, την ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τις παρεμβάσεις της σε καθοριστικά σημεία. Σαν παράδειγμα οι άδειε παραμονής, η διάρκεια των αδειών παραμονής, σαν καθοριστικό στοιχείο της σωστής διαδικασίας απορρόφησης. Εκτιμώ επίσης και τις προτάσεις που γίνονται για την εμπλοκή των τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων ευρύτερα υπέρ των προσφύγων. Η αξία των κοινωνικών υπηρεσιών που θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας ειδικά για τα μικρά παιδιά. Θα πρέπει επίσης να δούμε και τις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων, έτσι ώστε αυτοί που δικαιούνται διεθνούς προστασίας να έχουν εγγυημένη πρόσβαση και ταχύτατη στη δικαιοσύνη. Να ευχαριστήσω και την κυρία Ατζέα. Να πω ότι έχει και αυτή προσφέρει ιδιαίτερα στο κείμενο και δέχομαι τις προτάσεις της σαν παράδειγμα σχετικά με την βοήθεια η οποία γίνεται ε, για τους πρόσφυγες όχι μόνο γλωσσική μέσω διερμηνέων αλλά και μέσω διαμεσολαβητών. Επίσης σημασία έχει η κινητικότητα στο εσωτερικό ενός εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση και δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων των προσφύγων στο εσωτερικό της Ένωσης και επίσης ε, να μην αφήσουμε τις γειτονικέ χώρες να εκτίθενται τόσο πολύ και να φέρουν ε, στους ώμους τους μόνες το βάρος των φαινομένων αυτών. Απαιτούνται πόροι, απαιτείται τεχνική βοήθεια και θα πρέπει επίσης και μια ρύθμιση νομική που να θέσει τέλος στην διεστραμμένη λειτουργία της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε, για άλλες διευκρινήσεις. <coughs> Νομίζω ότι ήδη έχετε μελετήσει τις προτάσεις μου και είμαι πεπισμένος ότι και μετά από αυτά τα οποία σας είπα έχουν διαμορφωθεί τα θεμέλια για μια σωστή δουλειά και την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τον Τόμας Μάντορα θα πάρει το λόγο η κυρία Μωρά Ή κάποιος άλλος. Συμφωνήστε μεταξύ σας και πείτε μου. Ο Σορσμπαχ συνάδελφος ε, Τόμας Μαν με παρακάλεσε να παρουσιάσω την τοποθέτησή του γιατί δυστυχώ δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα στην Τσουριξέλα ε, γιατί είναι στο Βερολίνο όπου συμμετέχει σε μία διάλεξη. Επεξεργάστηκε την πρόταση ε, με τους συναδέλφους, το 1 τρίτο των τροπολογιών κατατέθηκε και από το ΕΛΚ. Αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για εμάς τους χριστιανοδημοκράτες και είναι ικανοποιητική η συμφωνία στις γενικότερες γραμμές. Επεξεργάστηκε τις 377 ε, τροπολογίες τις τελευταίες ημέρες και ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα. Θέλουμε από κοινού να φροντίσουμε για την κοινωνική ενσωμάτωση στο σημείο 8 καθώς και η αξιολόγηση των ε, επίσημων και ανεπίσημων ε, ικανοτήτων, οι γλωσσικές ικανότητες είναι σημαντικές και σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει στο 16 να αναφερθεί και τα σχετικά με το κοινωνικό ταμείο. Τονίζουμε τη σημασία των συνδικάτων, της ε, ε κοινωνίας των πολιτών στο σημείο 22 και αυτό που επίσης είναι πολύ απαραίτητο είναι οι τροπολογίε τη Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών, για την ιδιαίτερη κατάσταση των γυναικών και των παιδιών. Αλλά ο Τόμα Μαν πιστεύει ότι θα πρέπει να συζητηθούν και πολλά θέματα, γιατί θα πρέπει να τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο η οδηγία, προκειμένου τα άτομα τα οποία ζητούν τέτοια διεθνή προστασία αργότερο μετά από τι έξι μήνε να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία. Είναι πολύ φιλόδοξο αυτό, θεωρεί ο Τόμας Μάν στο σημείο 24 και επίσης το θέμα της επανένωσης των οικογενειών ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το θέμα των κατωτών μισθών. Ένα βασικό πρόβλημα είναι οι ορισμοί. Το βασικό πρόβλημα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ιδιαίτερα η σύγχυση που προκαλείται με τους όρους, γιατί στο σημείο 2 ο συνάδελφος Μπράντο ε, Μπραντ Μπενιφέη διαπιστώνει σωστά τις ε, συνθήκες που επικρατούν και η διάθεση συμβιβασμού καταδεικνύει ότι θα πρέπει να υπάρξουν σωστοί ορισμοί από όλες τις ομάδες, γιατί τα άτομα τα οποία μας απασχολούν Για τα άτομα αυτά, μάλλον στις 377 ε, χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι. Ε, ε, μετανάστες πρόσφυγες, άτομα τα οποία έχουν σκόπο να μείνουν, άτομα τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας, άτομα με καθεστώς πρόσφυγα και προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία των συμβιβασμών θα πρέπει να διευκρινίσουμε σύμφωνα με τον Τόμας Μαν ε, τους ορισμούς ποιον θέλουμε να έχει τέτοια πρόσβαση στους ε, κοινωνικούς μας, ε, στις αγορά εργασία, στις κοινωνικές μας δομές και το καθεξής. Όλοι, σας ευχαριστώ πολύ, η Έλικα Στίβενς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλημέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον εισηγητή γιατί τόσο καλή δουλειά που έχει κάνει. Το τελικό κείμενο είναι ισορροπημένο και καλά στοχευμένο. Βέβαια, έχω κάποια επικριτικά σχόλια να κάνω, οπότε επιτρέψτε μου. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπάρχει ένα πράγμα που να λέγεται «Η πρόσφυγες» διάβασα ότι έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στις ομάδες εκείνες προσφύγων που είναι πιο αδύναμες, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι κάθε πρόσφυγας είναι ένα άτομο που έχει το δικό του υπόβαθρο, τα δικά του προσόντα και τις δικές του ανάγκες. Σήμερα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ε, δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γυναίκες πρόσφυγες. Γι' αυτό προτιμάω μία προσέγγιση ένταξης εξατομικευμένη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις συγκεκριμένες προκλήσεις της κάθε ομάδας προσφύγων. Θα ήθελα επίσης στην έκθεση να δω πιο ξεκάθαρα να λέει ότι οι προσπάθειες ένταξης να γίνουν πιο πολύ για αυτούς οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα μείνουν περισσότερα χρόνια στην Ευρώπη. Δεν έχουμε αρκετούς πόρους, οπότε τα χρήματα πρέπει να δαπανώνται καλά. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας από τη μια τις διαδικασίες ε, ασύλου και την άλλη και απ' την άλλη την ένταξη των προσφύγων. Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι δεν πιστεύω πως οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο μπορούν να είναι η λύση για το πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη. Γι' αυτό δεν είναι η λύση η μπλε κάρτα. Ε, το προσφυγικό και το ασφαλιστικό είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το άσυλο δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη πρέπει να φροντίσουν να βρούνε τις κατάλληλες συνθήκες και οι προϋποθέσεις για απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Μόνο τότε εξάλλου θα ενταχθούν και καλύτερα οι πρόσφυγες στις κοινωνίες μας. Τέλος, πιστεύω ότι η ευελιξία στην αγορά εργασίας μπορεί να βοηθήσει πιο γρήγορα να ενταχθούν στις κοινωνίες μας οι πρόσφυγες. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του και πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ επικοδομητικές συναντήσεις των σχεδόν εισηγητών και προσλέπω σε καλή συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Ναι, η ευελιξία ενδεχομένω σε περιπτώσει να οδηγήσει και σε αντίθετα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα έξυπνο, ένα ευφυέ μήνυμα προς τα έξω, τόσο προς τους Ευρωπαίους πολίτες και προς όσους θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και τις δύο αυτές κατηγορίες ανθρώπων. Και στηρίζω τον εισηγητή για το έργο του. Είχα ήδη την ευκαιρία να κοιτάξω τις συμβαστικές τροπολογίες και είδα ότι πολλά από αυτά που η δικιά μου πολιτική ομάδα πιστεύει ότι είναι σημαντικά, συμπεριλαμβάνονται ήδη στις συμβαστικέ τροπολογίες. Ένα κοινό σύστημα ασύλου που θα βελτιώσει τις διαδικασίες αναγνώρισης. Ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρίες Δέστητες ε, πολιτικές όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας μια συνολική προσέγγιση επίσης όσον αφορά την κοινωνική ένταξη για να μην υπάρχουν πολλές πιθανότητες απομόνωσης να δώσουμε σημασία στην αναγνώριση των ήδη υπαρχόντων προσόντων και δεξιοτεχνιών των προσφύγων. Ένας μόνιμος μηχανισμός μετακατάστασης για όλες τις χώρες μέλη είναι το ελάχιστο δείγμα αλληλεγγύης που μπορούν να επιδείξουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δείξουν ότι συμμετέχουν σε μια ένωση και δεν πρόκειται για συσσόρευση χωρών. Όπως πολύ σωστά είπε και ο συγητής, υπάρχει τροπολογία που έχουμε υποβάλει για το ελάχιστο ή το ανώτατο όριο χρόνου για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας έξι μήνες το πολύ, λέει ο εισηγητή, αλλά γνωρίζουμε και από την παρουσίαση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι πολλές χώρες μέλη δίνουν λιγότερο χρονικό διάστημα. Φοβάμαι λοιπόν ότι αν πούμε έξι μήνες, αυτό μπορεί να πλήξει τη στάνταρτ πολιτική σε πολλές χώρες. Αν και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η πρόσβαση στην αγορά εργασίας όσο γίνεται πιο γρήγορα ακριβώς για να αποφεύγονται προβλήματα, να μην νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί ότι είναι στην απομόνωση. Πάντως, βρίσκω πολύ καλές αρκετές ιδέες που υπάρχουν στην έκθεση που επιμένει στην πρόσβαση, στην εκπαίδευση, στη στέγαση, στις υπηρεσίες. Όλα αυτά όντως συνεισφέρουν στην ορθή αποκατάσταση επαγγελματική των προσφύγων. Όντως και εγώ περιμένω τις ε, συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών και σίγουρα θα συνεργαστούμε πολύ καλά για να καταλήξουμε σε ένα ακόμα καλύτερο κείμενο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κονζάλης Πένας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενό του και τον ευχαριστώ και για τα σχόλιά του και όλα όσα μας είπε σήμερα. Είναι μια περίπλοκη βέβαια έκθεση αυτή. Υπάρχουν αντιφατικές ε, απόψεις μεταξύ μας, το βλέπουμε αυτό και με τις τροπολογίες. Οπότε ευχαριστώ για την προσπάθεια που έχει κάνει με τις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που μας έφτασαν χτες. Ελπίζω να στηριχτούν οι τροπολογίε εκείνε οι οποίε αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων, όλων των διακρίσεων και να στηριχτούν και τροπολογίε που έχουν κοινωνικό περιεχόμενο και αναφέρονται στην πρόσβαση στην υγεία, στην εκπαίδευση, την ε, κοινωνική προστασία ή τη στέγαση των ετούντων άσυλο και προσφύγων. Πρέπει εδώ το κράτος να κάνει περισσότερα το κάστοτε κράτος και κυρίως για όσους είναι πιο ευάλωτοι και απαιτούν διεθνή προστασία. Όσον αφορά την τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε και ο εισηγητής για τα επαγγελματικά προσόντα, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πιστεύουμε ότι είναι καλό να αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα, αλλά βέβαια ποτέ αυτό δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διακρίσεις όταν αποφασίζουμε για αιτήσει ασύλου. Επίσης, θέλω να αναφερθώ και στις ε, ξενοφοβικές ε, εκκλήσεις που ακούμε στην Ευρώπη, που για μας είναι παραφωνία. Τα σχόλια εκείνα δηλαδή, τα οποία θέλουν να δώσουν την εντύπωση ότι η ευθύνη μας για την απόδοση του καθεστώτος ασύλου πλήττει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και τη δικιά τους ευημερία. Είναι επικίνδυνος ένας τέτοιος λόγος, είναι λάθος. Το μόνο το οποίο φταίει και θέτει σε κίνδυνο τους πολίτες μας είναι η λιτότητα η οποία εφαρμόζεται κυρίως στις ε, χώρες που βρίσκονται στην Νότια Ευρώπη. Το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εξάλλου από το τεχνικό κλιμάκιο που έλεγε ότι αν δεν εφαρμοστούν τώρα μέτρα ένταξη στην αγορά εργασίας των προσφύγων, αμέσως ή μεσοπρόθεσμα, τότε μακροπρόθεσμα, αυτό θα σημαίνει πολύ μεγαλύτερο οικονομικό και πολιτικό κόστος και κόστος όσον αφορά τη συνογή στις κοινωνίες μας. Υπογραμμίζω λοιπόν το ατομικό δικαίωμα κάθε ατόμου προκειμένου να ζητήσει διεθνή προστασία και το δικαίωμα που έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας με έναν ελάχιστο μισθό και έχει δικαίωμα επίσης και στην οικογενειακή επανένωση. Άλλο σημαντικό στοιχείο για μας. Μόνο πολιτική βούληση χρειάζεται. Οι τροπολογίες που μπερδεύουν διάφορα θέματα και που ε, παριστάνουν ότι ε, προσφέρουν περισσότερα στους ετούντες άσυλο ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της ε, χώρας υποδοχής δεν έχουν νόημα εδώ. Ούτε και η προσπάθεια να θεωρηθούν εγκληματίες οι πρόσφυγες, ενώ ακριβώς αυτό που θέλουμε είναι να παλέψουμε εναντίον των συμμοριών. Σύμφωνο πάντως ότι χρειάζονται μηχανισμοί προκειμένου να βοηθήσουμε γρήγορα τους πρόσφυγες. Η υποδοχή των προσφύγων πρέπει να γίνεται έτσι όπως έχουν δεσμευτεί οι χώρες μέλη και να μειωθεί σε έξι μήνες το διάστημα μετά από το οποίο μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να έχουν άδεια εργασίας τα άτομα αυτά. Ελπίζω λοιπόν και εμείς και εγώ με τις ε, απόψεις μου να μπορώ να συνεισφέρω στο έργο του συγκητή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τζιν Λάμπερτς δεν είναι εδώ. Τζέρι. Εσείς. Η Λάουρα Ατζέα τότε είναι η επόμενη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συνάδελφο Μπενιφέη για την πρότασή του και για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε. Τον ευχαριστώ επίσης γιατί ήδη έχει κυκλοφορήσει τις πρώτες συμβιβαστικές τις οποίες επεξεργαζόμεθα και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται. Οι θέσεις τις οποίες του εκφράσαμε δεν ήταν πάρα πολλές, αλλά νομίζω ότι ήταν σημαντικές και κατεπίγουσες. Εμείς ζητήσαμε μια δίκαιη κατανομή των ευθυνών, έναν μηχανισμό υποχρεωτικής κατανομής δηλαδή των υποχρεώσεων στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Αυτά είναι μέτρα τα οποία μπορούν να γίνουν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλεγχος μεταναστευτικών ροών, να σταματήσουμε αυτούς που δεν έχουν ε, δικαίωμα εισόδου, να διακρίνουμε τις κατεπίγουσες δράσεις από ένα σχέδιο το οποίο να είναι μεσοπρόθεσμης περίοδου έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Να αξιολογήσουμε σωστά τις καταστάσεις που επικρατούν στις διάφορες χώρες που υποδέχονται τους πρόσφυγες και οι χώρες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις μεταναστευτικές ροές ε, σαν αντιστάθμισμα για τη μείωση του κόστους της εργασίας. Έχει λοιπόν σημασία να ε, δώσουμε εγγυήσει στους πρόσφυγες τη στιγμή που έρχονται στην Ευρώπη, να τους δώσουμε επίσης βοήθεια και ε, γλωσσική και νομικοί ε, και ε, πολιτιστικούς διαμεσολαβητές για να βοηθήσουμε την ενσωμάτωσή τους. Οι πολιτικές, ε, οι κατεπίγουσες στις οποίες υποχρεούμεθα να προσφεύγουμε δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας στην παρούσα φάση όπως ε, η ενδιάμεση αναθεώρηση του Ταμείου για το άσυλο και τα λοιπά που λόγω της κρίσης την οποία βιώνουμε έχουν ήδη εξαντληθεί οι πόροι στα μισά του χρόνου. Δώσαμε λοιπόν τρία δις στην Τουρκία για να βοηθήσουμε στην διαχείριση των μεταναστών. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει με αποτελεσματικό τρόπο να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέψει τα επόμενα χρόνια τα μεταναστευτικά ρεύματα να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά. Να επιταχύνουμε την επεξεργασία των αιτήσεων. Εδώ γίνεται και μία αναφορά νομίζω στην οδηγία μπλε κάρτας που σαν ιδέα είναι καλή αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας και οι προτάσεις μας. Εξετάζουμε τις συμβιβαστικές προτάσεις προς το παρόν και ευχαριστούμε τον συνάδελφο Μπενιφέ για μια εξαιρετικά περίπλοκη αλλά ευαίσθητη και κατεπίγουσα προσπάθεια. Είμαστε λοιπόν στην διάθεσή του για να προετοιμάσουμε ένα αποτελεσματικό έγγραφο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μιλάω αντί για την Jean Lamberts, λέει η κυρία Ρένκε, που δεν μπορεί να είναι εδώ. Εκ μέρου τη ομάδα μα, λοιπόν. Ε, μα ικανοποιεί πολύ η έκθεση και στηρίζουμε πολλέ από τι τροπολογίε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τι επικοδομητικέ του προτάσει. Κυρίω για τι τροπολογίε εκείνε που ενισχύουν το ρόλο των τοπικών αρχών και τη κοινωνία των πολιτών. Είναι ζωτική σημασία, διότι αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο μέσο στήριξης για να συμμετέχουν πραγματικά για το άσυλο και οι πρόσφυγες στην αγορά εργασίας. Ευχαριστούμε επίση και για το γεγονός ότι λάβατε υπόψη σας πολλές από τις τροπολογίες μας, εκείνες δηλαδή που κυρίως θέλουν να υπογραμμίσουν τις προσπάθειες που γίνονται για να αλλάξει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για μας αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι δεν μπορεί να κοιτάμε μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις. Πρέπει να δούμε πώς τους ετούντες άσυλο και τους πρόσφυγες μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε μακροπρόθεσμα στην αγορά εργασίας. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι πολλές δικές μας ε, τροπολογίες είναι καλό που έχουν ληφθεί υπόψη. Εξακολουθούμε βέβαια να συζητάμε το κατά πόσο πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ταμείο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αν δεν υπάρχουν επιπλέον χρήματα, τότε μπορεί να υπάρξει ανταγωνισμό ανάμεσα σε προγράμματα που ήδη υπάρχουν και που είναι πολύ χρήσιμα. Μιλάμε για περισσότερη ευελιξία. Εμείς στηρίζουμε αλλαγές επίσης στα πλαίσια των, των πολιτών δημοσιονομικών πλαισίων, ιδίως το σημείο 16. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και προσβλέπουμε και εμείς σε επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας. Πρόεδρος, Μαραπιτσότο. Πιτσότο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έπρεπε να έχουμε μία έκθεση για το θέμα των μεταναστών. Νομίζω ότι προσπαθούμε να καλύψουμε αυτή την έλλειψη από την άλλη είναι σαν αθλητική δραστηριότητα αυτό το οποίο κάνουμε. Βγάζουμε εκθέσεις αλλά πέραν αυτού η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Οπότε είναι προφανές ότι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε δεν είναι ο σωστός. Ελπίζω όμως ότι η Ευρώπη δεν θέλει να κάνει εισαγωγή χιλιάδων και εκατομμυρίων σκλάβων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελα να πω στον συνάδελφο Μπενιφέη το ότι το να υπερασπίζεται κανείς ε, τους πολίτες της χώρας του, τους συμπατριώτες του δεν είναι, ε, δεν είναι λάθος, δεν είναι έγκλημα. Εγώ αυτό κάνω. Και ο εισηγητής κάνει εδώ ένα λάθος. Μίλησε με τα συνδικάτα, μίλησε με τις ενώσεις των μεταναστών, με όλο τον κόσμο μίλησε, αλλά δεν μίλησε με τους ανέργους της πόλης του, της χώρας του. Το 40% των νέων στην Ιταλία δεν έχουν δουλειά. Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς αυτά τα παιδιά ότι ένας ε, μετανάστης έχει δικαίωμα στη δουλειά και αυτός όχι. Δεν ξέρω με τι λόγια θα το πει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της εργασίας καταρχάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι γίνονται πόλεμοι και ο κόσμος πεθαίνει, αλλά και στην Ιταλία πεθαίνει ο κόσμος από ανεργία. Υπάρχουν αυτοκτονίες και χθε στην περιοχή μου για κάποιον ο οποίος έχασε τη δουλειά του. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με περισσότερο ρεαλισμό. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστικό κόμμα, είμαστε ρεαλιστικό κόμμα. Εμείς απλά βλέπουμε πώς έχει η κατάσταση. Και γι' αυτό οι τροπολογίες μας δεν θα ήταν σωστό να τις εξετάσεις μόνο σου, αλλά να τις συγκρίνεις με την πραγματικότητα της ε, χώρας μας. Δεν είναι ρατσιστικές, είναι λογικές. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει πρώτα να καλύψουμε το πρόβλημα της ανεργίας στην Ιταλία. Και το θέμα δεν είναι να εισάγουμε εκατομμύρια σκλάβων, επαναλαμβάνω. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Αυτό το οποίο λέμε και το επαναλαμβάνουμε ότι το θέμα της μετανάστευσης πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στις χώρες προέλευσης. Θα πρέπει να ελέγχουμε τους ανθρώπους που έρχονται. Όταν φτάνουν στην Ιταλία εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και λιγότερα από το 30% παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα, αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κόβουν βόλτες στην Ιταλία παράνομα και οι άνθρωποι αυτοί ε, πολλές φορές ε, λειτουργούν εκτός νόμου και αποτελούν ένα πρόβλημα για την κοινωνία μας. Πρέπει λοιπόν στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούσετε με μεγαλύτερη προσοχή τα κόμματα αυτά, τα οποία αυτό το οποίο θέλουν είναι το θέμα της μετανάστευσης να τεθεί σε ένα πλαίσιο έλογο και τότε μόνο θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με παραγωγικό τρόπο. Γιατί αλλιώς θα είναι η έκθεσή σας μία ακόμα άχρηστη έκθεση. Δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο και γι' αυτό λοιπόν θα δώσω το λόγο στον Πράντον Μπενιφέη. <laughs> Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια από τα στοιχεία στην κυρία Μπιτζότο. Η έκθεση δεν αφορά τους μετανάστες, αλλά αφορά τους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο. Είναι διαφορετικό θέμα. Ε, δεν μιλάμε για εισαγωγή σκλάβων, αλλά το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, που μοιάζει πολύ στην δουλεία. Ε, το πρόβλημα της διάκρισης ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι ε, προέρχονται από καταστάσεις τρομερές έτσι ώστε να τους αναγνωριστεί η διεθνής προστασία είναι κάτι το διαφορετικό από την οικονομική μετανάστευση. Και αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με πραγματισμό και με ε, λογική όπως το αναγνωρίζουν όλες σχεδόν οι πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι πολλές φορές ε, η κοινή λογική βρίσκεται στη μεγάλη πλειοψηφία των θέσεων και γι' αυτό πρέπει να διαβάσετε η κυρία Μπιτζότο την έκθεση. Λέτε ότι δεν υπάρχει η επιθυμία να αποφύγουμε τους κινδύνους και θέλουμε να χτυπήσουμε άλλες κατηγορίες όπως οι νέοι άνεργοι μέσω της πολιτικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Μα αυτό κάνει η έκθεσή μου. Λέγω ότι η πολιτική ενσωμάτωση των μεταναστών, των προσφύγων μάλλον, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινωνικό ντάμπινγκ, δεν θα πρέπει να χειροτερεύσει τις συνθήκες εργασίας των αυτοκτόνων και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πιστώσεις της συνοχής μειώνοντας τις παροχές προς τις λιγότερο ευνοημένες κατηγορίες για να καλύψουμε τις ανάγκες των προσφύγων. Αντίθετα κυρία Μπιτζότο, εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί το κοινωνικό ταμείο για να καλύψει μια νέα κατάσταση η οποία δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εις βάρος των ασθενεστέρων κοινωνικά. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να κάνει επικοδομητικές προτάσεις και όχι σκέτη προπαγάνδα και με έξοδα μάλιστα του φορολογούμενου. Θα ήθελα επίσης να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί όπως είπαμε υπάρχει μια γυτνίαση των θέσεων της πολιτικής μου ομάδας και άλλων ομάδων, ιδιαίτερα στην ανάγκη ταχύτερης παρέμβασης, στην ανάγκη ενίσχυσης των ταμείων για την κοινωνική συνοχή, ενίσχυσης των διαδικασιών χορήγησης ασύλου, και ένα κοινό σύστημα λοιπόν. Υπάρχουν πολλά τα οποία μένει να γίνουν. Ε, υπάρχουν πολλές διαφορές, θα πρέπει να τις συζητήσουμε τις διαφορές αυτές με τους σκιώδεις συζητητές για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την ισορροπία ανάμεσα στην βελτίωση των δεξιοτήτων χωρίς διακρίσεις εις βάρος των ε, προσφύγων να προσπαθήσουμε επίσης να σταθμίσουμε σωστά τις ανάγκες κάθε κατηγορίας έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα μέσα παρέμβασής μας. Και εδώ τίθεται και το θέμα της χρηματοδότησης κυρίως, πάνω στο θέμα της χρηματοδότησης υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ μας. Έχω την αίσθηση όμως ότι μπορεί να υπάρξει μια πλειοψηφία έτσι ώστε όπως έχω προείπει να αποφύγουμε δράσεις που θα βοηθούν τους πρόσφυγες αλλά θα είναι εις βάρος άλλων κατηγοριών. Αυτό το αποκλείουμε. Θα πρέπει επίσης να, να διευκρινίσουμε πλήρως σε επίπεδο ορολογίας την παρέμβασή μας, σε ποιους απευθύνονται οι υπηρεσίες, σε ποιους, θα καλύπτει το κοινωνικό σύστημα και με ποιο τρόπο. Σε επίπεδο ορολογίας δηλαδή κάποιες διαφορές μεταξύ μας υπάρχουν και θα πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τους όρους. Κλείνοντας, φύγουμε όπως είπα και κάποια άλλα θέματα όπως τη στήριξη των τοπικών οργανώσεων, των τοπικών αρχών που ασχολούνται με τέτοια προβλήματα και την ανάγκη να υπάρξει και μια διαπολιτιστική παρέμβαση και πέραν αυτών όπως είπα υπάρχει μια κοινή αντίληψη για το πρόβλημα στις περισσότερες πολιτικές ομάδες Υπάρχουν στοιχεία δύσκολα βέβαια όπως η οδηγία για την μπλε κάρτα ε, όπου έχουν ακουστεί διαφορετικές απόψεις αλλά στα υπόλοιπα ε, υπάρχει μια συνένεση, υπάρχει μια κοινή βάση στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων Νομίζω ότι θα κλείσουμε την προσπάθεια αυτή με χρήσιμο τρόπο για την Ευρώπη, με χρήσιμο τρόπο για τους Ευρωπαίους πολίτες, έτσι ώστε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και σε νομοθετικό επίπεδο και να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να ενσωματώσουμε τους πρόσφυγες όχι εις βάρος άλλων κατηγοριών λιγότερο ευνοημένων. Ευχαριστώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ. Στις 30 Μαΐου θα ψηφίσουμε, Μαΐου θα ψηφίσουμε στην ε, ε, Επιτροπή και τον Ιούλιο θα το δούμε στην ολομέλη το θέμα. Μάλιστα. Και να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 8 της σημερινής διάταξη. Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου στην Ευρώπη. Είμαι εγώ εισηγητής. Μία ε, παρατήρηση να κάνω ευθύς εξ αρχής. Για το θέμα αυτό ήταν σαφές ότι υπήρχε πραγματικά ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον από πλευρά των μέλων τη Επιτροπή, αλλά το γεγονό ότι δέχτηκα 282 τροπολογίε μετά την πρώτη συζήτηση που κάναμε για το θέμα αυτό με εξέπληξε. Δεν θέλω να επισέλθω απαραίτητα σε... στις μεμονωμένες τροπολογίες και είναι και πάρα πολλέ. Σκοπός ε, της, ε, των τροπολογιών είναι να εμπλουτίσουν ασφαλώς το κείμενο και η πρώτη ομάδα των τροπολογιών ακριβώς αυτό το σκοπό έχει, να εμπλουτίσει και να συγκεκριμενοποιήσει την έκθεση αυτή. Αυτό λοιπόν είναι θετικό. και θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμβαστικές τροπολογίες. Η δεύτερη ομάδα τροπολογιών είναι βασικά γλωσσικής φύσεως και θεωρώ ότι αυτό μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με τη διευκρίνηση κάποιων ε, όρων στην έκθεση. Και σε αυτό θεωρώ ότι θα έχουμε προβλήματα στη συνεργασία μας με τους κοιοδείς. Η τρίτη ομάδα τροπολογιών είναι αρκετά αμφιλεγόμενες αν θέλετε, γιατί ουσιαστικά αυτό που λέτε θα πρέπει τα πράγματα να παραμένουν ως έχουν. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι εντάξει, μπορούμε να την αφήσουμε κατά μέρος αυτή την έκθεση, αλλά δεν είναι αυτό σκοπός και πρόθεσή μας, γιατί σε διάφορες τοποθετήσεις, ανακοινώσεις, έγγραφα της Επιτροπής ε, και του Κοινοβουλίου τάσσομεθα κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, υπέρ της συμμετοχής των ε, ατόμων, υπέρ της κοινωνικής δομής κτλ. Και θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ε, έχουμε ως στόχο το να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, γιατί θα έχουμε αποτύχειες προς την επίτευξη του στόχου μας. Η τέταρτη ομάδα τροπολογίων με μου προξένησε κάποια έκπληξη και πρέπει να σας ομολογήσω ότι με διασκέδασε κιόλα. 62 στον αριθμό τροπολογίες, οι οποίες θέλουν να διαγράψουν ολόκληρα τμήματα, ολόκληρες παραγράφους από την έκθεση αυτή. Αν ε, τις δεχτούμε, θα μείνουν μόνο οι επικεφαλίτες και 40% του περιεχομένου της έκθεσης. Και αυτό φαντάζομαι ότι δεν αποτελεί σκοπό του υπεύθυνου της κατάρτισης της έκθεσης στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, ταχθήκαμε κατά της ε, οδηγίας ε, ad personam και αυτό το απορρίψαμε με συντριπτική πλειοψηφία γιατί αυτή η οδηγία δημιουργεί τη δυνατότητα να παρακάμψει κανείς εθνικές προδιαγραφές, να τις, ε, μην τις σεβαστεί. Και αν θέλουμε λοιπόν να διαγραφούν αυτά τα κομμάτια, ουσιαστικά είμαστε αντίθετοι με τις λήψεις αποφάσεων ως τώρα της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Επίσης, ε, διαπιστώνουμε την ανάγκη να συμπληρωθεί το τοπίο σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν ως θέση προσπαθούμε να το βάλουμε εδώ και καιρό στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε λοιπόν δεν καταφέραμε να το πετύχουμε αυτό και τώρα αυτή θα ήταν μια καλή ευκαιρία να το να συμπεριλάβουμε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, παρατηρήσεις ε, για το κείμενο. Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή επιτάπητος δεν είναι ε, σοσιαλιστική διαβολική έκθεση και κανείς ε, δεν έχει την πρόθεση να αγνοήσει, να συνενώσει τα 28 διαφορετικά συστήματα. Υπάρχουν 28 διαφορετικά κρατημέλη και συμπεριλαμβάνεται και η Νορβηγία σε ό,τι αφορά τα, τη συμμετοχή στο Δυτικό Συμβούλιο. Κατά δεύτερον, καμία επιχείρηση δεν θα υποχρεωθεί να αλλάξει μορφή. Αυτό είναι απόφαση που λαμβάνει εθελούσια κάθε επιχείρηση, αν το λάβει ως απόφαση. Δεν είναι σκοπός μας να επιλέξει καθή, κανείς μόνο τις που του αρέσουν. Η έκθεση αυτή ζητά ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα σέβονται το ευρωπαϊκό δικαίου, αλλά θα πρέπει να τηρούνται κάποια ελάχιστα πρότυπα σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση εργαζομένων. Αυτός είναι ο στόχος ε, της έκθεσης. Φαντάζομαι ότι θα είναι συναρπαστική η συζήτηση για την έκθεση αυτή και θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή ο κ. Λάρε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, όπως είπα και στην πρώτη ομιλία για την έκθεση αυτή, το δικαίωμα πληροφόρησης και οι συμβουλές προς τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ζήτημα, γιατί αυτό μπορεί να προαγάγει την αποδοτικότητα. Οι εργαζόμενοι επίσης έχουν δικαίωμα σε αυτή την πληροφόρηση και στη σχετική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ορίζεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τα διάφορα εθνικά συστήματα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν υποδεικνύω τη σημασία της επικουρικότητας στις τροπολογίες μου. Ξέρουμε ότι το κάθε εθνικό σύστημα προέκυψε από την εθνική παράδοση και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε την Βέλγια, την Ιταλία, την Ολλανδία, σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή η παράδοση. Στο Μιλάνο, για παράδειγμα, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ρόλος σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, παρόλο που δεν υπάρχει σχετική παράδοση και θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να λεπτούν σχετικές πρωτοβουλίες. Διαπιστώνουμε επίσης ότι το ΕΛΚ δεν είναι υπέρ της ε, έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη νέων δεσμευτικών προδιαγραφών. Δεδομένη τη κατάσταση στα κράτη-μέλη, θεωρούμε ότι δεν είναι επίκαιρο κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε την εντύπωση, δεδομένη τη κατάσταση, ότι θα πρέπει να λεφτούν υπόψη και οι συγκεκριμένοι όροι. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την έκθεση πρωτοβουλία και προσβλέπω και εγώ στις μελλοντικές μας συνομιλίες και στις συναντήσεις με τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο κύριος Μαρτάν, πρώτα και μετά βρήκε. Για διαδικαστικό. Εγώ θέλω το λόγο. Λέει ο κύριος Καλβέ Σαμπό. Για διαδικαστικό, ναι. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά πρέπει να φύγω τώρα για ένα λεπτό σιγής μπροστά στο ημικύκλιο. Αν συμφωνείτε θα πάρω το λόγο αργότερα. Αλλιώς απλώς ζητώ συγγνώμη που πρέπει να αποχωρήσω, αλλά το καθήκον μου είναι αυτό. Είναι το μόνο που είχα να πω. Και ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τη διακοπή. Πρόεδρος. Καλώς. Θα επανέλθει. Θα γυρίσετε πάντως. Εντάξει, αφού θα επιστρέψετε, καλώς. Ωραία. Ματά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Εσάς δηλαδή. Η έκθεση αυτή πρέπει και πιστεύω ότι θα βοηθήσει υπέρ της κοινωνικής δημοκρατίας στις επιχειρήσεις. Εγώ, όπως το έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα, δεν θέλω να επιβάλλω το ένα σύστημα πάνω σε ένα άλλο. Φυσικά και πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις διαφορετικές συνήθειες και τις συνδικαλιστικές παραδόσεις. Το θέμα είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα γίνει αν προλαβαίνουμε τα προβλήματα, οπότε δρούμε έγκαιρα και αποφεύγουμε οικονομικά δράματα κοινωνική δημοκρατία. Σίγουρα στην Ευρώπη δίνονται πληροφορίες, αλλά όχι πάντα. Πολλές φορές τα πράγματα τα μαθαίνουμε από τον τύπο και τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι τα μαθαίνουν κατόπιν ορτής. Λοιπόν, αυτά που μας προτείνεις σίγουρα είναι μια καλή βάση προς συζήτηση. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες τροποποίησεις από την ομάδα μου για να μην επιβάλλουμε ένα μοντέλο πάνω σε ένα άλλο και κυρίως για να δώσουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενου, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις συνήθειες και τις παραδόσεις να είναι πιο αποτελεσματικοί και να επηρεάζουν πιο αποτελεσματικά τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Πράγματι πρέπει να υπογραμμίσουμε όλα τα θέματα γύρω από τη συμμετοχή, τη διαβούλευση κτλ ακόμα κι αν η συναπόφαση έχει δείξει στις βόρειες χώρες ότι είναι αποτελεσματική. Εγώ θα ήθελα αυτό να ισχύει παντού, αλλά βέβαια εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες των μεν και των δε. Για την επικουρικότητα και εμένα με ξέπληξαν κάποιες τροπολογίες. Εδώ δεν πρέπει να πούμε ότι μια αρμοδιότητα επιβάλλεται σε μια άλλη. Πάντως, είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχουν πολυεθνικές σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρόνως. Και έτσι φυσικά και θα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα οι εργαζόμενοι έτσι ώστε όχι να εναρμόσουμε την κοινωνική πολιτική, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα το ήθελα, αλλά αν μη τι άλλο να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε κάπως το επίπεδο των δικαιωμάτων αυτών που δεν έχουν αρκετά. Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα στην Ευρώπη σήμερα. Επιχειρήσεις δηλαδή πολυθρικές που δρούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρόνος. Τώρα η μονοπρόσωμη επιχείρηση, συμφωνώ με αυτό που λες. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Κάποιοι έχουν βρει τη χαραμάδα για να παρακάμπτουν κανόνες, οι εθνικές διαδικασίες όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση. Συμφωνώ με αυτά που είπες. Πρέπει να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα τάχιστα. Πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να έχουμε μια εναρμόνιση, συγχρόνως όμως να υπάρχει μια καλή διάρθρωση ανάμεσα στη συναπόφαση και την συμμετοχή, τη διαβούλευση Βασικά είναι η τροπολογία 167. Το κείμενο αυτό, εφόσον τροποποιηθεί καλά, μπορεί να βοηθήσει να ζήσει καλύτερη δημοκρατία προς το συμφέρον όλων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ατζέα. Πρόεδρε, ε, λέμε διάφορα ανέκδοτα μεταξύ μας, αλλά δυστυχώς ε, η έκθεση αυτή δεν παρουσιάζει τίποτα το αστείο. Όπως είδατε και από τις τροπολογίες που έχω καταθέσει, λέει ο κύριος Μπασίρ, εγώ και οι σκιώδεις συνάδελφοι, η πρόταση, οι, οι προτάσεις οι οποίες γίνονται είναι απαράδεκτες για πάρα πολλούς από εμά εδώ σήμερα. Από 282 τροπολογίες που κατετέθησαν, οι 61 προβλέπουν διαγραφές. Υπάρχει δυνατότητα επικοδομητικών τροπολογιών βέβαια και κάποιες είναι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία προτείνεται δεν είναι πολύ εφικτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ξεκινήσω με κάτι το θετικό. Υπάρχει μια αιτιολογική σκέψη την οποία στηρίζω. Το D κεφαλαίο. Λέγεται εδώ ότι η συμμετοχή και οι μορφές συμμετοχής των εργαζομένων σε επίπεδο διοίκησης επιχειρήσεων υπάρχουν σε 18 χώρες και στην Νορβηγία, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους σε επίπεδο ιστορικής και οικονομικής εξέλιξης και αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Μπορούν τα κράτη-μέλη ε, να μην παρεμβαίνουν στον τομέα αυτό. Φοβάμαι ότι όχι και οι διαφορές υποχρεωτικά είναι υψηλές. Κάθε οδηγία που θα προτείνεται θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες αυτές τις τεράστιες διαφορές και αυτό είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα γίνει. Η καταναμή των βέλτιστων πρακτικών θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε στο κόμμα των συντηρητικών. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες τις οποίες προτείνετε εσείς. Αυτή που, στην οποία εμένεται είναι ότι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να έχουν τις ίδιες εξουσίες με τους διαχειριστές. Ε, εσείς ε, που έχετε υπαλλήλους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτούς. Δεν νομίζω ότι θα τις στέλνατε να πάνε να ψηφίσουν για σας την Ολομέλεια και γιατί είναι κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους κανόνες για πολύ σωστούς λόγους. Δεν διαφωνώ ότι πρέπει να ακούσουμε τις απόψεις των εργαζομένων, κάτι το οποίο ε, θα βοηθήσει τους, ε, τη λειτουργία των εταιριών. Και εγώ σαν τέος ιδιοκτήτης επιχείρησης ε, θα έλεγα ότι αυτό έχει νόημα. Είναι καλό λοιπόν για τους εργαζομένους και την σωστή λειτουργία της επιχείρησης όμως έχουν υπάρξει, ε, υπάρχουν μάλλον οι διευθυντικές δομές μιας επιχείρησης για να πετύχει ε, φυσικά ε, τους στόχους της η επιχείρηση αυτή. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Εδώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει δικούς του κανόνες. Πάει μια χαρά χωρίς κανόνες και δεν θα ήθελε οι Βρυξέλλες ε, να πούνε στις επιχειρήσεις το Γιόξε το πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Οι προτάσεις εδώ διακανονισμού που γίνονται είναι το αντίθετο από αυτά τα οποία έχουν ανάγκη οι πολίτες μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, πιέζεται το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά να αποχωρήσει και οι τροπολογίες δείχνουν ότι δεν είμαι μόνος ο οποίος ε, ε, θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο, υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό το οποίο εσείς προτείνετε ουσιαστικά είναι το γερμανικό μοντέλο, το οποίο δεν ταιριάζει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ελπίζω στις συμβιβαστικές σας τροπολογίες να αλλάξετε τις προτάσεις σας έτσι ώστε να λάβετε υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες οι οποίες σήμερα εκφράζονται. So, Enrique noch nicht zurück, dann kommt Δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Ρίκε, ο ρίκε, η επόμενη ομιλητρέα. Ευχαριστώ. Και επιτρέψτε μου να διαφωνήσω έντονα με τον προλαλήσοντα. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς ε, μια συσσόρευση χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως καθήκον να ρυθμίζει κάποιους τομείς πολιτικής και το Ενωμένο Βασίλειο είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπροσώπηση των εργαζομένων δεν είναι σημαντική μόνο για να διασφαλίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και θέμα ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς. Γιατί αν ενισχύσουμε την ε, δημοκρατία, τότε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Βρετανοί πολίτες μπορούν να υποφεληθούν. Όταν διαβάζω λοιπόν την πρόταση αυτή, πιστεύω ότι κοιτάζοντα ανησυχίε για την επικουρικότητα, ή για διαφορετικές ε, συνήθειες και ανατροπίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τις ανησυχίες αυτές τις καθησυχάζει η πρόταση που εξετάζουμε. Παραμένουν οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο όταν πρόκειται για την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό το βήμα γιατί όπως είπα δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικών δικαιωμάτων είναι θέμα εσωτερικής αγοράς και δημοκρατίας τελικά. Αν λοιπόν κοιτάξουμε την πραγματικότητα βλέπουμε ότι για τις τιμές για παράδειγμα όπου εκπροσωπούνται καλύτερα οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις αυτές αντέχουν και πιο πολύ, είναι πιο ανθεκτικές. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει αυτή η πρόταση για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020. Πολύ σημαντικός στόχος για όλους μας. Η ομάδα μου λοιπόν στηρίζει την προσέγγιση αυτή, να έχουμε δεσμευτικούς και κοινού κανόνες όσον αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια και σε αυτό το επίπεδο, αν συνεργαζόμαστε και αν επικοδομητικά υπάρχει αυτή η συνεργασία των εργαζόμενων με τη δίκηση, τότε θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Θα μπορούμε να κοιτάμε ο ένας τον άλλον στα μάτια και να βρίσκουμε τις σωστές λύσεις. Και το τελευταίο, γιατί πιστεύω ότι οι τροπολογίες μας αυτό που προσπαθούν αυτό που προσπαθούν να υπογραμμίσουν, είναι ότι δεν είναι μόνο θέμα εργαζόμενων πώς θα συμμετέχουν σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων, αλλά επίσης πώς θα αντικατοπτρίζεται στις επιχειρήσεις και η διαφοροποίηση μεταξύ των εργαζομένων. Γι' αυτό μιλάμε για την ισότητα των φύλων και για την εκπροσώπηση κυρίως νέων, γιατί οι μαθητευόμενοι, οι εκπαιδευόμενοι στις επιχειρήσεις δεν ακούγονται όσο θα έπρεπε. Για μας θα ήταν μια σημαντική προσθήκη αυτή στις πολύ καλές προτάσεις που κατά τα άλλα έχουμε μπροστά μας από τον κύριο Χάντελ. Τέλος, με το προσωπικό μου, εγώ, έχω μια σχέση που κάθε άλλο παρά σχέση ιεραρχίας είναι. Και αυτό βοηθάει το κλίμα στο γραφείο μας. Και έτσι καταλήγουμε σε καλύτερες λύσεις για όλους. Οπότε από το πνεύμα αυτό, σαφώς και στηρίζουμε την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Τώρα η Λάουρα Ατζέα. Αλλά δεν είναι. ματά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή όλες τις μεγάλες ομιλίες που προηγήθηκαν και άκουσα και όλες τις υποσημειώσεις τις οποίες βάλατε σε αυτά που είπατε ότι εσείς κάνετε προτάσεις απλά και στόχος της έκθεσης είναι να υπάρξει μια ελάχιστη εκπροσώπηση των εργαζομένων και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις μεθοριακές επιχειρήσεις κτλ. Πάνω σε αυτή τη συζήτηση βέβαια οι απόψεις διαφέρουν. Πολλοί έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη. Εμείς πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι να συμμετέχουν στις λήψεις αποφάσεων. Φυσικά, γιατί πολύ συχνά στα εργαστήρια και στο χώρο εργασίας λύνονται τα προβλήματα. Όμως υπάρχουν αμφιβολίες για τις προτάσεις τις οποίες εσείς παρουσιάζετε σαν μη επιβαλόμενο πρότυπο. Το να ελέγχουν οι εργαζόμενοι τα διοικητικά συμβούλια δεν το δεχόμαστε. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είπε ο Εντουάβ Μαρτάν λίγο νωρίτερα. Είπε ότι εμείς θέλουμε να επηρεάσουμε τις στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων. Λέει δηλαδή το αντίθετο ακριβώς από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Θέλει λοιπόν να παρέμβει ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση ε, θα είναι όμοιρος των εργαζομένων. Ευτυχώς βέβαια αυτό αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές δεν φύγονται, αλλά αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση ιδιαίτερα όπου υπάρχει κρίση οικονομική. Ε, αυτά τα οποία επιθυμεί ο Εντουάρ Μαρτά του Μεγάλου Γαλλικού Συνδικάτου οδήγησε στην εξαφάνιση πολλών μεγάλων επιχειρήσεων ή στην μετακίνησή τους σε άλλες χώρες. Ε, και εκεί ευτυχώς που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα παρεμβεί, παρενεύει ήδη. Κλείνοντας λοιπόν, η παρέμβαση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εθνικό Δίκαιο στην ουσία βασίζεται σε μια πολύ υπερβολική ερμηνεία των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Και να πω στις φεμινίστριες φίλους, φίλες, το θέμα της ποσόστοσης των γυναικών δεν δικαιολογείται ούτε από την οικονομική αποτελεσματικότητα, ούτε από τις αρχές της αξιοκρατίας και της ίσης εκπροσώπησης. Θεωρώ ότι είναι υβριστικό για τις γυναίκες το να βάζουν με τέτοια ποσοστά. Υπάρχουν γυναίκες υπεύθυνοι μεγάλων επιχειρήσεων και δεν περίμεναν τις ποσοστώσεις για να προκόψουν. Ο κύριος Καλβέ Σομπον επέστρεψε Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και την κατανόησή σας. Και θα συνεχίσω στην Ισπανική. Για το συγκεκριμένο κείμενο, την πρόταση του Προέδρου, θα ήθελα να πω ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια είναι ένα σύμπτωμα των κοινωνιών που λειτουργούν με σωστό τρόπο και ένα χαρακτηριστικό των κοινωνιών που έχουν ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής ολοκλήρωσης και γι' αυτό συμμερίζομαι ε, την άποψή σας. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τρία βασικά θέματα τροπολογιών με τρεις βασικούς προσανατολισμούς που δεν είναι μόνο η δική μου προσωπική άποψη αλλά εκπροσωπούν και το σύνολο της πολιτικής μου ομάδας. Μετά από αυτά που ακούστηκαν θα ήθελα να σας παρηγορήσω ότι εμείς παρακολουθούμε ε, τις αλλαγές στον κόσμο αυτό και θα συμφωνήσουμε σε πολλά μαζί σας. Όμως σε τεχνικό επίπεδο το ένα εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια κτλ. Ο τίτλος εδώ δείχνει θα έλεγα ένα περιορισμένο τρόπο αντίληψης της ε, υπόθεσης αυτής Φυσικά και πρέπει να συμφωνήσουμε με το ότι εμείς είμαστε ένα νομοθετικό όργανο. Εμείς κάνουμε προτάσεις, ε, καταθέτουμε προτάσεις, καταθέτουμε γνωμοδοτήσεις. Εμείς δεν θεωρούμε και δεν πρέπει να θεωρούμε την συμμετοχή των εργαζομένων να συμμετέχουν στα συμβούλια τα διοικητικά με συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια πρότυπα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι θα πρέπει η συμμετοχή αυτή να γίνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και τι σημαίνει αυτό. Είναι προφανές ότι η συμμετοχή των εργαζομένων είναι κάτι το επιθυμητό και είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων που είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα ο πολιτισμός της κάθε χώρας, οι εμπειρίες της κάθε χώρας στον τομέα τον συνδικαλιστικό, στον τομέα τον επιχειρηματικό, ο ίδιος ο παραγωγικός ιστός. Υπάρχουν ιστοί παραγωγική μικροεπιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με τη χώρα. Ανάλογα με την ιστορία, με τον πολιτισμό για να μην πω και ανάλογα με το κλίμα της κάθε επιχείρησης. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τη νομική ιστορία του καθενός ε, και των δικαίων των εργαζομένων σε κάθε χώρα. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τις διαδικασίες αυτές, αλλά με ευφυή τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Και θα πρέπει επίσης να θυμίσουμε ότι αυτό το οποίο επιθυμούμε είναι να υπάρξει μια σωστή συμμετοχή των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν βάρος, θα πρέπει να έχουν άποψη, αλλά δεν θα πρέπει να συγχέεται αυτό με την διαχείριση των επιχειρήσεων, γιατί εκεί οι διαχειριστές είναι υπεύθυνοι. Έχει σημασία λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό, όχι μόνο για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση, αλλά επίσης ε, να ευαισθητοποιούνται τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι όταν τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Εδώ και 40 χρόνια είχαμε ζητήσει να γίνεται σωστή ενημέρωση, να ενημερώνουμε, να δίνουμε την πληροφορία, αλλά η ευθύνη για τη διαχείριση είναι στην επιχειρηματική ομάδα η οποία ελέγχει και διαχειρίζεται ακριβώς την επιχείρηση. Ο δεύτερος τομέας είναι οι προτάσεις διεκδικήσεις σχετικά με τις ισχύουσες οδηγίες για τη συμμετοχή των εργαζομένων. Τα λεγόμενα συνεργατικά μέσα, βελτιώνοντας τα μέσα τα οποία υπάρχουν. Τα πράγματα εξελίσσονται, πρέπει να επικαιροποιηθούν και να βελτιωθούν στους τομείς όπου τα πράγματα πάνε καλά απλά. Τι μπορεί να κάνει εδώ η Ευρώπη η Ευρώπη μπορεί φυσικά να κάνει συστάσεις, η Ευρώπη μπορεί να κάνει το λεγόμενο benchmarking, μπορεί να βοηθήσει, να δείξει πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα σαν πολιτική ομάδα σχετικά με το πού φτάνει η πιθανή νομική βάση που θα επέτρεπε μια άμεση παρέμβαση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκεκριμένα στα θέματα της ε, συμμετοχής στη διαχείριση των εργαζομένων. Νομίζω ότι αν επιμείνουμε σε αυτό τότε θα αποδυναμώσουμε τους στόχους που έχουμε μπροστά μας. Και η τρίτη ομάδα θεμάτων είναι αυτή η ιδέα ακριβώς που θα μας επιτρέψει η νομική βάση με συγκεκριμένο τρόπο και εμείς εδώ έχουμε μια κάποια απόσταση. Είπαμε ότι δεν μπορούμε σε πάρα, ε, σε πάρα πολλά σημεία να προχωρήσουμε αν δεν υπάρχει νομική βάση που το επιτρέπει. Αυτό το οποίο έχει σημασία να δούμε είναι αν αυτό το οποίο επιθυμούμε με την οδηγία αυτή να διασφαλίσουμε ένα δικαίωμα κάτι το οποίο μου φαίνεται ε, θεμελιώδες, δηλαδή συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά όργανα, ε, την, ε, σαν παράλλημα την λειτουργία των συνεργατικών επιχειρήσεων κτλ. Θα πρέπει να κάνουμε καθολικό το σεβασμό της αρχής αυτής. Θα πρέπει επίσης να δούμε ακριβώς ε, αν στόχος μας είναι να ε, γίνουν σεβαστά κάποια ελάχιστα επίπεδα ή θέλουμε να παρέμβουμε μέσω συγκεκριμένων οδηγιών ε, και να επιβάλλουμε απόψεις οι οποίες δεν είναι θα έλεγα καθολικές στην Ευρώπη αλλά εκπροσωπούν ένα και μόνο συγκεκριμένο πρότυπο. Συγγνώμη, Ενρίκε, δεν ήταν πολιτική αυτή η παρέμβαση, ήταν ε, θέμα χρόνου. Μετά από 7,5 λεπτά ομιλία. Δεν ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Θα κάνω και εγώ λοιπόν τι παρατηρήσει μου καταληκτικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του ε, συναδέλφου, αλλά να σα παρακαλέσω, σα παρακαλώ όλου, να διαβάσετε. Να διαβάσετε. Αν δεν διαβάζετε, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Γιατί πολλά από αυτά που διατείνεστε. Δεν τα λέει καν η έκθεση. Το πρώτο θέμα του κυρίου Σαμπον. Του κυρίου Σαμπον. Κοιτάξτε, είμαστε σε επίπεδο ε, έκθεσης σε ό,τι αφορά την ανάθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη κάποια μέτρα στις επιχειρήσεις στο μέλλον. Κατά δεύτερον, η έκθεση αναφέρει ρητά το σχέδιο έκθεσης μάλλον ότι το δικαίωμα διαχείρισης της, ε, διαχείρισης της κυβέρνησης δεν αμφισβητείται κατά τρίτον. Αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα δεν ε, δεσμεύουν για τίποτα. Αν ληφθούν υπόψη, το θέμα δεν είναι συνάδελφέ μου, να υπερισχύσει το ένα μοντέλο του άλλου. Όχι, μιλάμε για ελάχιστα πρότυπα, τα οποία δεν έχουν σκοπό να αμφισβητήσουν το εθνικό δίκαιο, αλλά... Επιτρέψτε μου κύριε Μπασίρ, στην Ευρώπη δεν είναι εφικτό να ακολουθούμε αυτό το μοτίβο, γιατί στους τομείς, σε κάποιους άλλους τομείς με την ίδια λογική θα έπρεπε να αναστείλουμε τις εργασίες μας και παλιά δεν υπήρχαν και ευρωπαϊκά ε, διοικητικά συμβούλια, ε, βγάλαμε μία οδηγία με κοινέ προσπάθειε και των τριών θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε. Ε, αν το θέμα λοιπόν είναι κάθε φορά να βγαίνουμε και να λέμε ότι σε θέματα εργασιακού δικαίου δεν είναι εφικτό τίποτα, ε, τότε τι θα κάνουμε. Τίποτα. Αλλά αν υπάρχει μια ευρωπαϊκή ε, νομική ένα ευρωπαϊκό νομικό περιεχόμενο και ε, αυτό το περιεχόμενο ε, επιτρέπει να εφαρμόζονται καλύτερα το εθνικό και τοπικό και περιφερειακό δίκαιο, θα πρέπει να λυθούν όλα αυτά υπόψη. Υπάρχουν τα πικουρικά συστήματα αλλά δεν θέλουμε να εκμεταλλεύεται κανείς τα κοινά τα παρεφράκια που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο για να τα χρησιμοποιεί κατά των εργαζομένων. Κανείς δεν θέλει να εφαρμόσει οποιαδήποτε μορφή, για παράδειγμα, ε, διαχείριση στους Βέλγους, στο Βέλγιο, αν το θέλουν οι ίδιοι οι Βέλγοι. Αν δεν ε, συνάδει αυτό με την πολιτισμική, οικονομική, κοινωνική παράδοση του Βελγίου. Δεν τίθεται λοιπόν αυτό το ζήτημα της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης και συνδιαχείρισης. Αλλά αν ληφθούν ε, αποφάσεις, όταν λαμβάνονται αποφάσεις, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται. Αυτό είναι καθήκον μας ως Επιτροπή Απασχόλησης και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιαστεί η συζήτηση σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή και απλώς βλέπω στη συζήτηση αυτή στις 15 Ιουνίου θα κατατεθεί η έκθεση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ελπίζω να υπάρχουν κάποιοι καλοί συμβιβασμοί μέχρι τότε, οι οποίοι και να συγκεντρώσουν την υποστήριξη της πλειοψηφίας. Και νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο διελεύκανσης του τι εννοείται με την έκθεση αυτή μεταξύ των σκιωδών. Θα έχουμε άλλους δύο γύρους συζητήσεων, θα καταρτήσουμε τις συμβαστικές μας προτάσεις και θα δούμε πόσο μακριά θα φτάσουμε με αυτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι ολοκληρώσαμε και την ημερήσια διάταξη για το σημερινό πρωινό. Θα τα ξαναπούμε στις 3 με τις ψηφοφορίε Καλό διάλειμμα και καλή όρεξη.